Ja, ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen, die heute den Weg hierher gefunden haben und die Tagesordnung. Όσον αφορά την ημερήσια διάταξη, μπορούμε να τη δεχτούμε όπως ε, έχει, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, καμία παρατήρηση, οπότε την εγκρίνουμε ως έχει. Περνάμε στο σημείο 2 όλες οι γλώσσες εκτός από τα κροατικά, εκτός από τα μαλτέζικα και τα εστονικά είναι διαθέσιμα σε αυτή τη συνεδρίαση. Και περνάμε στον τριμερή διάλογο, έκθεση Παναγιώτοφ, που θα λάβει η χώρα η δεύτερη φάση τον Ιούνιο. Η προηγούμενη συνάντηση ήταν τέλος Απριλίου. Αύριο θα έχουμε 48 προσκεκλημένους, η Ντάκμα Ροτμπέρετ από το Βερολίνο. Αύριο θα τους φέρει και θα τους φυσικά χαιρετήσουμε και επισήμως αύριο. Αύριο έχουμε το εργαστήριο από τις 12.30 ως τις 3.30 αύριο στις 12.30 με 3.30 στην ε, αίθουσα PAS 5 Β1. Και περνάω στα πρακτικά του Ιανουαρίου 23-24, Φεβρουαρίου 25 και 26 εγκρίνονται χωρίς παρατηρήσεις. Περνάω στο τέταρτο σημείο της σημερινής διάταξης. Είναι η έκθεση του συναδέλφου Ζανόνη. Και σας δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα ξεκινάμε την πορεία της αναθεώρησης ε, της ε, οδηγίας ε, ΕΠΕ για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το 2011 του 1992 θεωρώ ότι η αναθεώρηση αυτής της οδηγίας είναι πολύ σημαντική, διότι η οδηγία αυτή είναι πολύ σημαντική για την ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι πάρα πολλά τα ε, προγράμματα τα οποία πρέπει να τύχουν αξιολόγηση εκδικτύπου, όπως για παράδειγμα ε, αεροδρόμια, ε, ε, εκμεταλλεύσεις εντατικής καλλιέργειας πουλερικών και θα πρέπει να γίνεται μία δημόσια ε, ή ένα ιδιωτικό έργο πριν ε, δοθεί η έγκριση, αν θεωρηθεί ότι υπάρχουν επιπτώσεις για το περιβάλλον, θα πρέπει να υποβάλλεται και σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ως διαδικασία θα πρέπει τα έργα τα οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας να είναι βιώσιμα από πλευράς περιβαλλοντικής. Η οδηγία χωρίζει τα ε, έργα αυτά σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Αυτά που προβλέπονται από το παράρτημα 1, τα οποία πάντα υπόκεινται σε διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως για παράδειγμα πυρηνική σταθμή, αυτοκινητόδρομο και το καθεξής, και αυτά τα οποία εμπίπτουν στο παράρτημα 2, που έχουν ίσως ε, λιγότερες επιπτώσεις, για παράδειγμα χιονοδρομικά κέντρα, τα οποία θα πρέπει ε, να υποβάλλονται σε εκτίμηση επιπτώσεων αναπερίπτωση. Υπάρχει η λεγόμενη διαδικασία screening δηλαδή και εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους αναδόχους και οι αρμόδιες αρχές ε, και θα πρέπει να βλέπουμε και τι ε, συμμετοχή θα πρέπει να έχει ο δημόσιος τομέας στη διαδικασία λήψης ε, αποφάσεων. Στα 28 χρόνια που εφαρμόζεται η οδηγία αυτή, διότι η πρώτη οδηγία εφαρμόστηκε το 1985, έγιναν τρεις τροποποίησεις, ενώ το πολιτικό, γεωγραφικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλάζει συστηματικά. Επίσης ε, υπάρχουν κάποια νομικά προσκόμματα, ε, υπήρξαν κάποιες προσαγωγές στο δικαστήριο και Μόνο στην οδηγία για τους φυσικούς οικοτόπους είχαμε λίγο λιγότερες ε, προσφυγές στο δικαστήριο. Γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μία τροποποίηση της οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη καταρχάς τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεύτερον, Κάποιου νέου πολιτικού στόχου που αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω για παράδειγμα την αποτελεσματική χρήση των πόρων, την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο, τη βιοπικιλότητα και την προστασία του περιβάλλοντο εν γέννη. Και οι βασικέ τροποποίησει που περιλαμβάνονται στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καταρχά η διαδικασία επαλήθευση για να δούμε κατά πόσον υπόκεινται στην οδηγία τα έργα, ε, να γίνεται επίση το λεγόμενο scooping, τρίτον να καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα και να λαμβάνονται κατά κατάλληλε αποφάσεις και τέταρτον να απλουστευτεί η διαδικασία. Ας δούμε λίγο τη διαδικασία επαλήθευση την οποία αποκαλούμε screening. Σε αυτή τη διαδικασία για να δούμε αν θα πρέπει να κάποια έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2 να τύχουν αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα δεύτερο παράρτημα, 2α, όπου ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει μία σειρά από συγκεκριμένε πληροφορίες στην αρμόδια αρχή, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία της ε, εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα ζητάται όταν θα υπάρχει ουσιαστική ε, επίπτωση για το περιβάλλον και να μην ζητάμε εκτίμηση επιπτώσεων όταν δεν θεωρείται απαραίτητο. Όταν ζητάμε συγκεκριμένε ε, πληροφορίες ε, θα εξοικονομούμε χρήματα και δεν θα υπάρχουν αμφισημίες και έτσι δεν θα ζητάτε από εκεί και πέρα από την αρμόδια αρχή ε, να ε, συμπεριλαμβάνει την εκτίμηση επιπτώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης διεύρυνε και τα κριτήρια επιλογής τα οποία προβλέπονται στο παράρτημα 3 και καθόρισε ότι η αρμόδια αρχή θα πρέπει να αποφασίζει εντός τριών μηνών ή το αργότερο εντός έξι μηνών εάν ένα πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται στο παράρτημα 2 θα πρέπει να έχει και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεύτερον, η ποιότητα των πληροφοριών της ε, εκτίμησης επιπτώσεων. Για να βελτιωθεί υπόψη, η ποιότητα, συγγνώμη, εισάγεται η διαδικασία scoping, που σημαίνει ότι καθορίζουμε ε, τι επίπεδο λεπτομέρειας θα έχουμε στην ε, περιβαλλοντική έκθεση. Να υπενθυμίσω ότι η περιβαλλοντική έκθεση είναι το πιο σημαντικό έγγραφο το οποίο θα αποτελέσει βάση ανάλυσης για τα κατά πόσον θα εκδοθεί ή όχι έγκριση για ένα συγκεκριμένο έργο για να μπορέσει η αρμόδια αρχή να λάβει συγκεκριμένε αποφάσει με το παράρτημα 4, έχουν συμπεριληφθεί οι πληροφορίε που θα πρέπει να δώσει ο ανάδοχο ε, στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λαμβάνοντα υπόψη καταρχά την υποχρεωτική αξιολόγηση των λογικών εναλλακτικών λέσεων που έχουν ίσω μικρότερη περιβαλλοντική επίπτωση. Δεύτερον, να βλέπει τι γίνεται και αν υπάρχει παρακολούθηση μετά την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ε, αν υπάρχουν ε, πολύ σημαντικέ αρνητικέ συνέπειε για το περιβάλλον, τρίτον πληροφορίε για τη βιοπικιλότητα, χρήση φυσικών πόρων, αλλαγή του κλίματο και κίνδυνο φυσικών καταστροφών. Ε, η τρίτη μεγάλη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος για τη λήψη απόφασης και η απλούστευση της διαδικασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει χρονοδιάγραμμα για να γίνει ε, διαβούλευση ε, εντός 30 ή 60 ημερών μέχρι κατεξαίρεση 90 ημέρες. Κατόπιν, το χρονοδιάγραμμα για τελική απόφαση είναι τρει μήνες και υπάρχει δυνατότητα παράτασης ε, στους έξι μήνες και τέλο υπάρχει και μια συντονιστική αρχή ε, μια μορφής ε, one-stop shop, μια ενιαία θηρίδα, στην οποία θα μπορούμε να αποφθούνται οι ανάδοχοι για την εκτίμηση περιβαλλοντικών υποπτήσεων μαζί με οποιαδήποτε άλλη αξιολόγηση μπορεί να ζητήσουν ε, οι αρμόδιες αρχές, ε, όπως για παράδειγμα ε, στοιχεία για την οδηγία για τις εκπομπές, διοξιδίου του άνθρακα, για τους φυσικούς σκοτόπους και το καθεξής. Τώρα, ποιε είναι οι δικέ μου προτάσει σε αυτό το σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την πρόταση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξάνει πολύ σημαντικά το επίπεδο της ισχύωση οδηγίας, γι' αυτό και ακριβώς εγώ υποστηρίζω αυτό το σχέδιο οδηγίας, το οποίο θεωρώ ότι είναι καλό. Έχω κάνει μια σειρά από προτάσεις τροπολογίας, οι οποίες στόχο έχουν να ενισχύσουν αποκλειστικά και μόνο την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλουμε να έχουμε και κάποια στοιχεία για να είναι πιο αποτελεσματική, χωρίς ε, να αλλάξει σε καμία περίπτωση η τοποθέτηση του συγκεκριμένου σχεδίου οδηγίες πρότεινα 61 τροπολογίες που αφορούν κυρίως καταρχάν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία λήψης απόφασης. Δεύτερον, να περιορίσουμε το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Τρίτον, να προβλέψουμε διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση ε, εκ των υστέρων ελέγχων που θα αποδείξουν ότι υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον. Τέταρτον, να πλουστεύσουμε ε, τη διαδικασία υποβολής ε, και επαλήθευσης της ε, περιβαλλοντικής έκθεσης. Πέμπτον, ασφάλεια δικαίου. Και έκτον, να συμπεριλάβουμε στο παράρτημα 1 προγράμματα για μη συμβατικά καύσιμα, όπως για παράδειγμα το σχιστολιστικό φυσικό αέριο. Όσον αφορά τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε μεγαλύτερο βαθμό, θέλει να ενισχυθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων και λαμβάνοντας υπόψη τη σύμβαση του άρχους πιο συγκεκριμένα στη διαδικασία του screening ε, και στην παρακολούθηση και στην περίπτωση που τα κράτη-μέλη αποφασίσουν να ανατρέξουν στις παρεκκλήσεις που προβλέπονται στη συγκεκριμένη οδηγία. Όσο περισσότερο συμμετέχει το κοινό και οι τοπικές αρχές, όπως για παράδειγμα η Δήμη, τόσο μειώνεται ο κίνδυνος ε, να υπάρχουν σημαντικές ε, δυσκολίες από νομική και προσφυγές στο δικαστήριο όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις στα κράτη-μέλη. Ε, δεύτερον, πρέπει να αποφύγουμε το μεγάλο πρόβλημα τη σύγκρουση συμφερόντων. Στην Ιταλία διαπίστωσα ότι παρά το γεγονό ότι υπάρχει επίσημο διαχωρισμό μεταξύ αρμόδια αρχή και αναδόχου, ε, Ιδίω όταν είναι όμως δημόσιο πρόσωπο ανάδεχο, ε, πολλές φορές συμβαίνει να υπάρχει ε, επιρροή μεταξύ των δύο και αυτό φυσικά υποσκάπτει την όλη διαδικασία και φυσικά και την ε, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατά την άποψή μου λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι θα υπάρχει απόλυτη ανεξαρτησία μεταξύ αρμόδιας αρχής και αναδόχου ώστε να μην υπάρχει και διαφθορά. Τρίτον, θα πρέπει να προβλέψουμε και συλλογικέ δράσεις για την εκ των υστέρων παρακολούθηση η οποία θα μας ε, οδηγήσει σε διαπιστώσεις ε, για αρνητικέ συνέπειες για το περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ε, προτείνω όταν υπάρχουν προβλήματα και συνέπειες για το περιβάλλον θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα. Εάν τα μέτρα λοιπόν είναι αποτελεσματικά δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά αν είναι μη αποτελεσματικά, τότε θα πρέπει να βρεθούν κάποιες λύσεις και σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει, ε, να λάβει διορθωτικά μέτρα για να διορθώσει τις ζημίες που προκαλούνται στο περιβάλλον. Τέταρτον, θα πρέπει να πλουστεύσουμε τη διαδικασία ε, ε κατάρτισης και επαλήθευσης της εκθέσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή... Ε, πρότεινε για να υπάρχει συγκεκριμένο αριθμό εμπειρογνωμόνων που κάνουν την αξιολόγηση, να υπάρχει ένα κατάλογο συγκεκριμένων ε, εμπειρογνωμόνων. Επειδή όμω είναι πολύ αυξημένο το στόχο για του αναδόχου και για τα κράτη-μέλη, θεώρησε ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη και στου αναδόχου αυτή την υποχρεωτική διαδικασία διαβούλευση με εμπειρογνώμονε. Οι εμπειρογνώμονε αυτοί μπορεί να είναι πολύ σημαντικά άτομα σε ακαδημαϊκό και πανεπιστημιακό επίπεδο και που μπορεί να μην ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό και εδώ διαφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει όμως, εάν υπάρχουν αυτοί οι πυρογνώμονες, να είναι απόλυτα ανεξάρτητοι σε θέματα περιβάλλοντος. Είτε είναι αυτοί οι οποίοι ε, καταρτίζουν την έκθεση επιπτώσεων, είτε συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή που θα πρέπει να ελέγξει την έκθεση από πλευράς τοπικών αρχών. Ασφάλεια δικαίου τώρα. Για να μπορέσουμε να έχουμε την κατάλληλη ασφάλεια δικαίου, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής ορισμός για τη βιοποκυλότητα βάση ε, της ε, Σύμβασης Όνου για την βιολογική βιοποικιλότητα. Υπάρχει μία αναδρομική εφαρμογή της οδηγίας ε, σε κάποιο σημείο, γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές σημείο αναφοράς για τις αρμόδιες αρχές και για τους αναδόχους, διότι υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει αλλά να μην έχουν περατώσει ακόμα την ε, επαχτή διαδικασία της αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε περίπτωση λοιπόν που έχει προχωρήσει κάποιο έργο και έχει ήδη κατατεθεί η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά την άποψή μου θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ε, χρησιμοποιώντας την παρούσα οδηγία. Επίσης, το πρώτο παράρτημα θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και τα μη συμβατικά καύσιμα, όπως για παράδειγμα το σχιστολευτικό φυσικό αέριο. Αυτό το ζήτησα και στην πράξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα... Ε, του 2012 για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ε, για τις διαδικασίες εξόριξης πετρελαίου ε, φυσικού αερίου και σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σε αυτό το ε, ψήφισμα ζητήθηκε να συμπεριληφθεί στο παράρτημα της οδηγίας και η κατηγορία των μη συμβατικών υδρογοναρθράκων έτσι ώστε τα διερευνητικά προγράμματα και τα προγράμματα εξόριξης να έχουν υποχρεωτικά και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τέλος, έχω συμπεριλάβει και μια σειρά από δευτερεύουσες τροπολογίες διότι θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνδράμει τα κράτη-μέλη ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τη διαδικασία του one-stop-shop. Να υπάρχει μια ενιαία θηρίδα, μια αρμόδια αρχή, η οποία θα συντονίζει τις υπόλοιπες αρχές, ώστε να μπορούν να εκδίδουν και όλες τις υπόλοιπες ε, εκτιμήσεις επιπτώσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου. Επιπλέον, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προβλέπουν αποτελεσματικές κυρώσεις, ε, ε, βάση και της οδηγίας αλλά και των εθνικών τους ε, νομοθεσιών. Μέτρα τα οποία θα αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την εφαρμογή προβληματικών πρακτικών. Και επίσης όσον αφορά τη διαδικασία του salami slicing, δηλαδή το να ε, κομματιάζει κάποιος, να διαιρεί ένα έργο να κόβει ένα έργο σε πολλά κομματάκια ώστε να φαίνεται ότι είναι μικρότερη επίπτωση για το περιβάλλον, αυτό θα πρέπει να το ε, αποφύγουμε με κάθε τρόπο. Θεωρώ λοιπόν ότι η συγκεκριμένη οδηγία και η τροποποίηση της οδηγίας θα σημαίνει ότι θα περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις ε, σημαντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα και να δούμε πόσο αποτελεσματική είναι η χρήση των πόρων μας, η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και να μην χάνουμε βιοπικιλότητα. Θεωρώ λοιπόν, χάρη και στην πολύτιμη συνεισφορά των μελών ε, της Επιτροπής μας, θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε ένα πολύ στεναρό κείμενο τον Ιούλιο, το οποίο θα συμμερίζονται αρκετοί. Θα ακούσαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον την άποψη των σχεδόν εισηγητών, των άλλων συναδέλφων και φυσικά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο. Είναι πολύ σημαντικό βεβαίως να αντιμετωπίσουμε εδώ τις προκλήσεις του 20 ου αιώνα και όσον αφορά διάφορες ε, εναλλακτικές λύσεις, ε, σχιστολιτικά αέρια και άλλες περιπτώσεις που σήμερα η Επιτροπή αντιμετωπίζει με έναν τρόπο μάλλον ε, επιφυλακτικό, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα εξετάσουμε. Η κυρία Γκροστέτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κριστίνα Γκουστιέρες δεν μπορεί σήμερα να είναι παρούσα. Μου ζήτησε λοιπόν να πάρω το λόγο εξ ονόματός της κάτι που κάνω ευχαρίστω. Αναγνωρίζει η κυρία Κουτιέρα ότι πρόκειται για μια πολύ καλή πρόταση. Θεωρεί όμως ότι δεν δίνονται λύσεις σε όλα τα σημεία τα οποία πολλές φορές παραμένουν ανοιχτά. Θεωρείται ότι Πρόκειται για θέματα που άπτονται των ε, περισσότερων ε, σημαντικών ε, τεχνικών θα έλεγα θεμάτων και η οδηγία σαφώς και θα πρέπει εδώ να βρει λύσεις για όλα τα εκρεμή σημεία. Αν κοιτάξει κανείς το σκεπτικό του κειμένου, διαβάζει ότι υπάρχει πολλή γραφειοκρατία, ότι υπάρχουν πολλά και διαφορετικά κριτήρια και ότι επιμηκύνονται οι διαδικασίες. Άρα χρειάζεται προφανώς απλοποίηση των διαδικασιών και σε εθνικό αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο. Η διοικητική πλευρά των διαδικασιών, η ε, έγκριση πολλές φορές είναι εξαιρετικά δύσκολη και μακροχρόνια και εδώ θα πρέπει να βρούμε τρόπους να γίνουν πιο γνωστά τα διάφορα σχέδια, να γίνεται η αξιολόγηση αντικτύπου και κάποια από τα σχέδια να μην περνάνε από την μελέτη αντικτύπου παραδείγματος χάρη όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Πρέπει να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά με αυτές τις διαδικασίες και θα πρέπει την ίδια ώρα όσον αφορά τις αρμοδιότητες να δούμε πώς θα μειώσουμε τη νομική ανασφάλεια γιατί βλέπουμε να ισχύουν πολλές φορές διαφορετικά κριτήρια από το ένα κράτος μέρος στο άλλο στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας. Δεύτερον, η κυρία Γκουτιέρες λέει επίσης ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ε, προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των διαφόρων τοπίων που πρέπει να προστατευθούν, αφού προηγουμένως περάσει και γίνει δεκτή και πιστοποιηθεί η διαδικασία αυτών των ε, επιπτώσεων του τοπίου. Πρόκειται για μία, αν θέλετε, προστασία του πολιτιστικού, αστικού περιβάλλοντος και κληρονομιάς, αλλά και του τοπίου. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε έναν κατάλογο που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα κράτη-μέλη όταν ξεκινούν μία ε, μελέτη αντικτύπου και αυτή, αν θέλετε, να γίνεται βάση των ίδιων κριτηρίων σε όλα τα κράτη-μέλη. Να αποτελέσει δηλαδή ένα είδος καταλόγου ή οδηγού που θα ισχύει και θα εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες, όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτό βεβαίως την οδηγία για τους ε, διαφορετικούς ε, οικότοπους, κάτι που θα πρέπει να καθορίσει προστατευμένες περιοχές και ζώνες, όπως ορίζει αυτή η οδηγία, είτε άλλες περιοχές, άλλες ζώνες που δεν ε, εποφελούνται από απολύτως καμία τέτοιου είδους προστασία. Αυτό προτείνει η κυρία Γκουτιέρες. Ελπίζω να παρουσίασα με ολοκληρωμένο τρόπο όλα αυτά που ήθελα να σας πει η κυρία Κουτιέρας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κρόστετ. Ο Πάβελ Μπρόκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του συναδέλφου μου Κρήτονα θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή συνεργασία την οποία είχανε, για την πολύ καλή προσέγγιση που έχει στο ζήτημα αυτό. Η οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να καταφέρουμε να αξιολογήσουμε σωστά οποιοδήποτε έργο ιδιωτικό ή δημόσιο μπορεί να έχει επιπτώσει στο περιβάλλον. Όλα τα έργα πρέπει, τα σχέδια έργων μάλλον, να εξεταστούν ακριβώ με κάθε λεπτομέρεια προτού υλοποιηθούν. Βέβαια είδαμε ότι υπάρχουν κάποιε αδυναμίες, κάποια κενά όσον αφορά την εφαρμογή στα κράτη-μέλη τη οδηγία αυτή και κάποιε επικαλύψει. Εμείς θα θέλαμε λοιπόν να καταφέρουμε να καλύψουμε τα κενά αυτά στην εφαρμογή, να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες στη δικασία του ελέγχου και να καταφέρουμε να κάνουμε τη σωστή ανάλυση όλων των έργων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να φέρονται επίσης και τα εναλλακτικέ προτάσεις στα σχέδια αυτά και θα πρέπει να προβλέπονται και περαιτέρω μέτρα ανακοφιστικά ή αντιστάθμισης ε, κάθε φορά που προβλέπονται σημαντικές σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θα πρέπει κάθε φορά βέβαια οι ανάδοχοι του έργου να αιτιολογούν και τη συγκεκριμένη απόφαση που λαμβάνεται για ένα έργο. Όσον αφορά την βιοπικιλότητα, τις κλιματικές αλλαγές θα πρέπει πάλι να προβλέπονται έργα για να μέτρα με συγχωρείτε ώστε να αποφεύγονται οποιαδήποτε αρνητικές, οποιασδήποτε αρνητικές επιπτώσεις να υπάρχουν για το περιβάλλον. Επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο περισσότερη συμμετοχή του κοινού σε όλα τα επίπεδα συνεργασίας σύμφωνα με τη σύμβαση του Άρχους. Θεωρούμε ότι το κοινό θα πρέπει να τυχαίνει διαβούλευση προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση πριν να αρχίσει τη διαδικασία screening, η διαδικασία scoping. Επίσης, συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα όπου η μετα... η υστέρων παρακολούθηση αποδεικνύει τελικά ότι υπάρχουν αρνητικέ επιπτώσει για το περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μία συνένεση στα πλαίσια των μέτρων ανακούφιση και αντιστάθμιση. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 φαίνεται ότι υπάρχει μια περαιτέρω δυνατότητα παρέκκλησης. Η εφαρμογή των παρεκκλήσεων της παραγράφου 3 και 4 θα πρέπει να την χάνουν ενός συστήματος περαιτέρω εγγυήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θα πρέπει να, να μας απομακρύνουν από την εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Στα πλαίσια της διαφάνειας θα θέλουμε στο άρθρο 6 να έχουμε ένα κοινό σημείο επαφή σε κάθε κράτος μέλος, έτσι ώστε να συμφωνούμε τελικά με το άρθρο 7 της οδηγίας, η οποία ήδη ισχύει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Τζανόνι για την έκθεσή του, για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε στα πλαίσια της αναθεώρησης οδηγίας για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα ήθελα όμως να τον ευχαριστήσω και να τον συγχαρώ για την ουσία, για το περιεχόμενο της εργασίας τους, καθώς, καθώς επίσης και τις τροπολογίες οι οποίες μας προτείνει, οι οποίες θεωρώ ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και θα ήθελα να τον διαβεβαιώσω ότι η δική μου πολιτική ομάδα των οικολόγων πρασίνων πραγματικά υποστηρίζει την προσέγγιση αυτή. Ο κύριος Ζανώνη το είπε ότι η οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει ως στόχο να ενδυναμώσει το σύστημα αξιολόγησης προκειμένου να καταφέρουμε, και αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε κάθε φορά, και να προλάβουμε τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάποιων έργων, να μειώσουμε τις επιπτώσεις αυτές, να τις καταργήσουμε και εντελώς. Στη χειρότερη των περιπτώσεων να αντισταθμίσουμε τις επιπτώσεις αυτές και να καταφέρουμε κατά κάποιο τρόπο, και αυτό υπόθηκε, να κάνουμε μια σωστή επιλογή ανάμεσα στα έργα εκείνα, τα οποία τελικά θα είναι λιγότερο αρνητικά για το περιβάλλον. Αν τώρα πραγματικά θέλουμε και αυτός νομίζω ότι είναι ο στόχος όλων των προτάσεων που έχουν υποβληθεί αν θέλουμε να ενδυναμώσουμε αυτή την, αυτές τις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις, τότε θα πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε, να συνδυάσουμε περισσότερο όλες τις τομιακές μας πολιτικές, προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να εφαρμόσουμε όλα τα νομοθετήματα τα οποία έχουμε εγκρίνει κατά τη διάρκεια της θητείας μας είτε πρόκειται για στόχους που έχουν να κάνουν με την στρατηγική για την καταπολέμηση της απώλειας βιοπικιλότητας, είτε πρόκειται για τη στρατηγική για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, είτε πρόκειται για, τον, για την έκθεση εκείνη την οποία εγκρίναμε πέρυσι όσον αφορά τη διατήρηση των υδάτων. Εγκρίνουμε λοιπόν και υποστηρίζουμε και την έκθεση και τις τροπολογίες του κ. Τζανόνη, ιδίως όσον αφορά επτά σημεία στα οποία θα αναφερθώ και τα οποία κατά την άποψή μας δεν θα πρέπει να αποδυναμωθούν σε καμία περίπτωση στην πρόταση την οποία έχουμε μπροστά μας. Από τη μια νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το να έχουμε στα πλαίσια των περιβαλλοντικών εκτιμήσεων ενός έργου τις επιπτώσεις στην βιοπικιλότητα και τις επιπτώσεις όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να προσθέσουμε και κάτι ακόμα, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ζήτημα του εδάφους. και προκειμένου να έχουμε μια πιο σφαιρική και όχι τομεακή προσέγγιση, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει και μια ανεξαρτησία των υπερογνωμόνων, προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε μια περιβαλλοντική εκτίμηση η οποία δεν θα βάλεται από σύγκρουση συμφερόντων. Και ως προς αυτό προτείνουμε μια διαδικασία πιστοποίησης ευρωπαϊκή και εθνική, Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω και θα μπορέσουμε να φερθούμε και στους διάφορους εκείνους οργανισμούς οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν αυτές τις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν τελικά και τους εμπειρογνώμονες και να πιστοποιήσουν ανεξαρτησία των εκθέσεων. Επίσης, υποστηρίζουμε την αναθεώρηση του παραρτήματος 1, καθώς επίσης και τη ρητή αναφορά που γίνεται στην εκμετάλλευση του συστολιθικού φυσικού αερίου, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο ακόμα και να αφαιρθούμε και σε αυτές τις δραστηριότητες αλλά και σε άλλες και να μην περιορίσουμε τελικά την αξιολόγηση σε συγκεκριμένα κατόφλια, αλλά να έχουμε μια περιβαλλοντική εκτίμηση η οποία θα καλύπτει μόνο την εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου, αλλά και την έρευνα για σχιστολιθικό φυσικό αέριο. και για άλλες νέες πηγές ενέργειας. Όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες τις οποίες ε, εμείς θα υποστηρίξουμε, θα ήθελα να σας πω ακόμα ότι ο εισηγητής ε, μας προτείνει ένα ενισχυμένο σύστημα υποχρεώσεων όσον αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων για ένα έργο. Και μας λέει ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται εναλλακτικέ αυτές προτάσεις, οι οποίες ε, μπορούν τελικά να μας οδηγήσουν στο να επιλέξουμε το πιο φιλικό προς το περιβάλλον έργο. Εμείς προτείνουμε να υπάρχει και μια ενισχυμένη πρόσβαση στο δικαστήριο, στα δικαστήρια, καθώς επίσης και μια πιο ενισχυμένη συμμετοχή των ε, ενδιαφερομένων, του κοινού. Όσον αφορά τώρα τη συντόμευση των δικαστικών διαδικασιών, εμείς θεωρούμε ότι όσο πιο σοβαρή και διαφανής τελικά είναι μια διαδικασία έγκρισης μάλλον και όσο περισσότερο συμμετέχει τελικά το κοινό, τόσο λιγότερες είναι και οι νομικές αντιπαραθέσεις οι οποίες προκύπτουν. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το επιχείρημα αυτό και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα έργα τα επαξιολόγηση θα ακολουθούν όλες τις νομοθεσίες και όλους τους σχετικούς κανόνες. Ολοκληρώνω τέλος λέγοντας και το ακόλουθο, πρέπει να γίνεται απαραίτητη διασύνδεση ανάμεσα στο να γίνονται αυτές οι περιβαλλοντικές εκτιμήσεις με τρόπο ενισχυμένο και ότι προφανώς αποφελείται και το κοινό από αυτό το πράγμα, εμείς προτείνουμε να υπάρχει και δυνατότητα αναστολής ή διακοπής των έργων ή να μην ξεκινάνε καν τα έργα αν υπάρχει μια νομική αντιπαράθεση και αν αποδεικνύεται τελικά ότι η περιβαλλοντική επίπτωση δεν είναι πλήρης, ότι δεν είναι επαρκής. Ολοκληρώνω τέλος ε, λέγοντας ότι όντως ε, η όλη αυτή οδηγία είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην πρώτη φάση ενός απότερου σχεδίου, το οποίο θα μας επιτρέψει να λάβουμε τελικά μία πλήρη πολιτική απόφαση. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερα στι πληροφορίε εκείνε οι οποίε μπορούν να μα κάνουν να αποδεχθούμε ένα έργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η πρώτη αυτή φάση στην έγκριση ενό έργου, η αξιολόγηση δηλαδή του έργου, να δυναμωθεί περισσότερο. Θεωρώ λοιπόν θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο την έκθεση αυτή του κυρίου Τζανόνι, που πραγματικά λαμβάνει υπόψη του πολύ περισσότερο από την υφιστάμενη νομοθεσία τι περιβαλλοντικέ μα ανησυχίε. Ευχαριστώ πολύ. Ο παίρνει Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα ECR χαιρετίζει την προσπάθεια να μειωθούν εδώ κάποιες άσκοπες ε, διαδικασίες τροποποιώντας αυτή την οδηγία. Θεωρούμε πραγματικά ότι ο εισηγητής έκανε εξαιρετική εργασία, είναι σαφέστατη η κατεύθυνση που επιλέγει. Παρ' όλα αυτά η ομάδα μας πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα έτσι ώστε να υπάρξει ισορροπία μεταξύ προστασίας του περιβάλλοντος και επιβολής ε, εμποδίων και ε, γραφειοκρατικού βάρους από τις αρμόδιες ε, αρχές. Εδώ μπορεί παραδείγματος χάρη να αυξηθεί και το κόστος ε, και ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών, κάτι το οποίο πρέπει να το αποφύγουμε. Και την ίδια ώρα να μην προστατευτεί περισσότερο το περιβάλλον. Θεωρούμε πραγματικά ότι και τα κράτη-μέλη και όλες οι αρχές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλα αυτά, ιδιαίτερα σε μια κρίση που προσπαθούμε να βγούμε από την οικονομική, σε μια περίοδο που προσπαθούμε να βγούμε από την οικονομική κρίση η εναρμόνιση για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντική από τη στιγμή που θέλουμε να επιβάλλουμε κοινά κριτήρια. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίσουμε τις ε, τοπικές αρχές, τις εθνικές αρχές να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν σε κάποιες τοπικές ιδιαιτερότητες. Όσον αφορά την ε, πρόταση για μία μοναδική θηρίδα, θα πρέπει εδώ να δούμε κατά πόσο αυτό εξυπηρετεί και διευκολύνει τον πολίτη. Θα πρέπει επίσης να δούμε ότι αυτές οι διαδικασίες πιστοποίησης πολλές φορές δημιουργούν μεγάλες γραφειοκρατικές δυσκολίες και για τα κράτη-μέλη ε, και για κάποιους αρμόδιους φορείς. Θα πρέπει να δούμε πώς εδώ αυτές οι διαδικασίες θα βελτιωθούν μειώνοντας τα εμπόδια και οδηγώντας προς περισσότερη ανάπτυξη. Θέλουμε να προωθήσουμε διαδικασίες για τις οποίες οι τοπικές αρχές είναι αρμόδιες για την επιλογή των πιο ικανών φορέων για να αναλάβουν ένα έργο. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα πρέπει να καλούνται, να ελέγχουν και να απελευθεύουν τις διαδικασίες και η επαλήθευση των στοιχείων και των πληροφοριών θα πρέπει να είναι επιστημονικά αντικειμενική χωρίς να υπάρχουν άλλου είδους επιρροές. Υπάρχουν κάποιες ασάφειες ακόμα σε αυτές τις προτάσεις και εδώ κινδυνεύουμε να βρεθούμε μπροστά σε μια νομική ανασφάλεια. Θα πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποια σημεία και να υπάρξει μια πιο σαφής διατύπωση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σιμάνσκι. Ο κύριος Σιμάνσκι. Zaproponowanie rozwiązań e, w załączniku <clears throat> na temat poszukiwania. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι υπερβολή να συμπεριλάβουμε κριτήρια επιλογής ε, στο παράρτημα όπως είχαμε αποφασίσει τον Νοέμβριο πέρσι, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να υπάρχουν πιο εκριβείς επιστημονικές πληροφορίες για το σκιστολιθικό φυσικό αέριο, θα μπορούσαμε να λαμβάνουμε μόνο αυτές τις πληροφορίες όταν ε, ξεκινά η διαδικασία. Και θεωρώ ότι τα κριτήρια αυτά μπορούν να αποτελέσουν πολύ σημαντικό πρόσκομα στη διαδικασία, ακόμα και αν έχουμε τις καλύτερες προθέσεις η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν θα πρέπει να αποτελεί ανάχωμα στην εξόριξη και την έρευνα για το σχιστολιστικό φυσικό αέριο. Οι πληροφορίες που διαθέτουμε μέχρι τούδε ε, καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ε, στο περιβάλλον ε, σε σχέση με την εξόριξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου και την εξόριξη φυσικού αερίου να σας παραπέμψω και στο ψήφισμα το οποίο εγκρίναμε στα τέλη του περασμένου έτους. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα ρυθμίσεων για την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Το σχιστολιθικό φυσικό αερίο θα πρέπει να υπόκειται στα ίδια κριτήρια επιλογής, τα οποία θεωρώ ότι ήδη διασφαλίζουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ακριβεί στο συγκεκριμένο έγγραφο, διότι η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ σημαντική. Δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, αλλά και την ε, ε, ενεργειακή, ε, την ασφάλεια σχεδιασμού ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ρίχα Σέμπερ είναι ο επόμενο. ομιλητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια καλή πρόταση σε γενικέ γραμμέ. Βεβαίω ε, πρέπει να μπούμε και στις διάφορες λεπτομέρειες. Άρθρο 2, όταν μιλάμε για το One Stop Shop, τη μοναδική θηρίδα. Εδώ θα πρέπει πραγματικά να δούμε ποιε είναι οι αρμόδιες αρχές και πώς θα καταφέρουμε να καθορίσουμε και να υιοθετήσουμε μία ενιαία διαδικασία οποία να ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη. Ποιε θα είναι οι αρμόδιε αρχές, παραδείγματο χάρη υπάρχουν ομοσπονδιακά κράτη, κράτη με διαφορετικέ δομέ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα γίνει η κατανομή των αρμοδιοτήτων και πώς οι διάφορες αρχές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο θα αναλάβουν. Καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχουν κάποιες συμβατικές ε, ε, υποχρεώσεις οι οποίες κινδυνεύουν να αντιμετωπιστούν με τελείω διαφορετικό τρόπο και να μην υπάρχει ενιαία διαδικασία τελικά στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν διάφορε προκλήσει και κίνδυνοι Γι' αυτό και ζητώ και εγώ πιο σαφείς ορισμούς έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να κατανοήσουν τι ακριβώς εννοούμε παραδείγματο χάρη όταν μιλούμε για υπηρεσίες, για οικοσύστημα, ένα οικοσύστημα παραδείγματο χάρη και οι παρεχόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια του οικοσυστήματος μπορεί να ερμηνευθούν με τελείως διαφορετικό τρόπο στη Βουλγαρία και στη χώρα μου. Άρθρο 4. Αναφέρουμε τις ε, ανάγκες και εδώ. Και εδώ οι διάφορες αρχές ε, των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν μια σαφέστατη περιγραφή του σχεδίου και το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι ποια είναι η σωστή διαδικασία. Συνήθως ουσιαστικά σε τέτοιες περιπτώσεις, πριν φτάσουμε στην αδειοδότηση, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες φάσεις. Εδώ έχω την εντύπωση ότι δεν περιγράφουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας και κινδυνεύουμε να βρεθούμε με επιπλέον εμπόδια και όσον αφορά το άρθρο 5, το επόμενο άρθρο και το scoping, εδώ επιβάλλεται μια επιπλέον υποχρέωση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι ακριβώς εννοούμε υποχρέωση, σε ποια φάση του σχεδίου εμπίπτει, για να δούμε αν αργότερα η διαδικασία διοδότησης ε, θα γίνει με τον αναμενόμενο τρόπο. Πολλά πράγματα δεν είναι πολύ ξεκάθαρα εδώ. Επίσης, όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες, Σήμερα η κάθε χώρα έχει ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί σε σχέση με τον ορισμό παραδείγματος χάνει των ε, εμπειρογνωμόνων. Υπάρχουν κάποιοι εμπειρογνώμονες, κάποιοι ειδικοί για όλες αυτές τις διαδικασίες. Το θέμα είναι ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν την πιστοποίηση. Άρθρο 8. Η διαδικασία διοδότηση. Πάρα πολύ σημαντικό άρθρο αυτό. Εδώ δεν περιγράφονται πολύ συγκεκριμένα κριτήρια στα οποία μπορούν να βασιστούν οι αρχές για το αν πρέπει ναι ή όχι να δοθεί η άδεια για ένα πρόγραμμα, για ένα σχέδιο. Οι αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, ναι. Αλλά εδώ υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη νομική ασάφεια για μένα. Πρέπει να καθοριστεί πολύ σαφέστερα το άρθρο 8 και τι ακριβώς εννοούμε για θετικά και αρνητικά σημεία. Κάτι άλλο που δεν μου φαίνεται ξεκάθαρο είναι οι προθεσμίες που δίνονται. Παραδείγματος τώρα για ένα μεγάλο αεροδρόμιο δεν είναι δυνατόν το τρίμηνο που ορίζεται εδώ να είναι αρκετό. Έχω την εντύπωση ότι εδώ αφήνουμε ένα τεράστιο περιθώριο Εκτίμηση και ερμηνεία στα κράτη-μέλη. Πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές όταν θέτουμε τέτοια κριτήρια και τέτοιες προθεσμίες. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Good afternoon. Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που δίνετε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πω ότι είναι χαρά μας που είμαστε εδώ και ευχαριστούμε ιδιαίτερο τον κύριο Τζανόνι για την εκθεσή του. Θεωρώ και εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ καλό το σχέδιο έκθεσης και σε μεγάλο βαθμό υποστηρίζει πλήρως και μεσθένος την έκθεσή μας και αυτό ε, κατά την άποψή μας είναι πολύ θετικό παρακολούθησα και τη συζήτηση και τα σχόλια των ε, υπολείπων μελών ε, της Επιτροπής και διαπιστώνω ότι σε πολλά σημεία υποστηρίζουν και αυτή την πρότασή μας. Σαφώ και υπάρχουν σημεία τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι η συνήθις ε, δημοκρατική διαδικασία. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι και η πλειονότητα των ενδιαφερομένων με τους οποίους διαβιλωθήκαμε κατά την προετοιμασία της πρότασης μας ε, συμφωνεί ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστεί η οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών υποπτώσεων και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και όλα τα διδάγματα τα οποία αντλήσαμε τα τελευταία 25 χρόνια στα οποία εφαρμόζεται η οδηγία αυτή. Αυτό ήταν και το συμπέρασμα της ευρεία ε, δημόσιας διαβούλευσης και οι αρχές οι οποίες διέπουν την αναθεώρηση, την αναθεώρηση και όπως ε, κατέδειξε και η δημόσια διαβούλευση, στόχο έχουν να ε, βελτιώσουν ε, τις ελλείψεις του παρελθόντος, αλλά να λάβουν υπόψη τους και τις κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις και να ε, ευθυγραμμίσουμε την οδηγία αυτή με την ευφυή νομοθεσία. Θα επανέλθω σε αυτό αργότερα, το ακούσαμε και από τους προηγούμενους ομιλητές και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία εξέδωσε αποφάσεις τα τελευταία χρόνια για τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών υποπτώσεων. Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα τα οποία περιλαμβάνονται στην πρότασή μας, ε, θα ήθελα να υπενθυμίσω τους δύο βασικούς στόχους που είχαμε όταν ε, ξεκίνησε η αναθεώρηση της οδηγίας. Καταρχάς, θέλουμε να βελτιωθεί η ποιότητα της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διότι όπως θα ακούσαμε και ήδη σήμερα από τα σχόλια, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, προκειμένου να διασφαλίσουμε ο μόνον ότι εφαρμόζουμε πιστά το περιβαλλοντικό δίκαιο που έχουμε στα διάφορα ε, σημεία της νομοθεσίας μας, αλλά για να έχουμε και τα ε, συνοδά υπόλοιπα ωφέλη που μπορούμε να έχουμε από την περιβαλλοντική νομοθεσία, ε, οικονομικές και κοινωνικές θετικές επιπτώσεις. Και τρίτον, θέλουμε η διαδικασία αυτή της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων να είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Αυτό και πάλι το αποκαλούμε εξορθολογισμό. Θα επανέλθω σε αυτό. Ε, είναι κάτι το οποίο ανησυχεί πολλούς από εσά εδώ στην αίθουσα. Θεωρούμε επίσης, ε, καθώς ακούσαμε και τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο, ότι πολλοί από τους στόχους τους οποίους ε, προσπαθούμε να επιτύχουμε είναι κοινοί. Αυτό το είδαμε και από τη συζήτηση προσανατολισμού που έγινε στο περιθάριο του Συμβουλίου ε, Υπουργών Περιβάλλοντος και ε, εκεί διαπιστώσαμε ότι πολλά από τα κράτη-μέλη καλωσορίζουν την πρότασή μας. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι δύο στόχοι που ανέφερα είναι αλληλένδετοι Χρειαζόμαστε καλύτερη ποιότητα, η οποία θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της οδηγίας και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεισφέρει και σε ίσους όρους ανταγωνισμού ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Και φυσικά ο εξορθολογισμός της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα βελτιώσει και την εφαρμογή της οδηγίας. Διάβασα πολύ προσεκτικά την έκθεση του κ. Τζανόνη και έχουμε ομαδοποιήσει τις τροπολογίες σε τρεις κατηγορίες και θα ήθελα να σας ε, κάνω μια σύντομη παρουσίαση, όχι πλήρη, των θεμάτων που εξετάσαμε. Καταρχάς υπάρχει μια κατηγορία στην οποία θεωρούμε ότι όντως ε, χρειάζεται περισσότερη βελτίωση και ενίσχυση της πρότασής μας και επειδή ακριβώς ο στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τους στόχους μας, θα ήθελα να ε, αναφερθώ στην τροπολογία 20 ή και στην τροπολογία 40 που αφορά την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, ε, τα οποία θα πρέπει να διατίθενται και στο κοινό. Επίσης, καλωσορίζουμε ιδιαίτερα και τις τροπολογίες, τις αιτιολογικές σκέψεις ε, για ε, κατεπίγουσα περιστατικά, ε, κατεπήγοντα περιστατικά, την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων. Όλα αυτά διέπουν φυσικά και τους λόγους για τους οποίους αποφασίσαμε να αναθεωρήσουμε την οδηγία και γι' αυτό ακριβώς και προτείναμε την αναθεώρηση. Μια δεύτερη κατηγορία τροπολογιών περιλαμβάνει τροπολογίες που ε, έκανε ο εισηγητής με στόχο ε, με να καλύψουν τους στόχους της πρότασης, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω το κείμενο όπως το προτείνεται. Παραδείγματο χάρη το θέμα τη ε, διαπίστευση των εμπειρογνωμόνων που προτείνει ο εισηγητή, τροπολογίε 28 έω 32 και λέει ότι θα πρέπει να καταργηθεί αυτή η διαδικασία. Και θα ήθελα εδώ ε, να σας υπενθυμίσω την ε, αξιολόγηση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καταδεικνύει ότι είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά αυτού του συστήματος. Υπάρχει σε αρκετά κράτη-μέλη και έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας πολύ καλός μηχανισμός παρακολούθησης της ποιότητας. Ταυτόχρονα ε, υπάρχει υποχρέωση για έλεγχο ποιότητας και εμείς είπαμε, και αυτό είναι σαφές στην πρότασή μας, ότι η επιλογή ενός μηχανισμού και ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί επαφίεται στα κράτη-μέλη. Επομένως υπάρχει περιθώριο ε, τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν πώς ακριβώς θα εφαρμόσουν το συγκεκριμένο μηχανισμό. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συζητήσουμε περαιτέρω τον καλύτερο δυνατό μηχανισμό, αλλά δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι μία από τις ε, ελλείψεις της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει έλεγχος ποιότητας και πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Αν δεν κάνω λάθος από αυτά που άκουσα και από τα σχόλιά σας, αυτό ε, επιθυμούν και πολλοί από όσους σχολίασαν το θέμα και ενδιαφέρονται επίσης και για την ανεξαρτησία αυτών που θα εξετάζουν τις ε, εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ένα άλλο παράδειγμα στο οποίο θεωρούμε ότι θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω κάποια θέματα είναι οι τροπολογίες που αφορούν τη συμμετοχή του κοινού στα διάφορα στάδια της διαδικασίας της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εμείς θεωρούμε ότι η πρότασή μας είναι και γνωρίζουμε ότι είναι βάση των στόχων της Σύμβασης του Άρχους για πρόσβαση σε πληροφορίες, δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία λήψης απόφασης και δεν θα πρέπει να λησμονούμε και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα περιβαλλοντικά μέτρα και γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στην Σύμβαση του Άρχους να σας πω ότι η παρούσα οδηγία περιλαμβάνει αρκετές διατάξεις που διασφαλίζουν κατάλληλη συμμετοχή του κοινού και των ενδιαφερομένων, παραδείγματο χάρη περιβαλλοντικές αρχές και δήμους και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει συμπεριλάβει και επιπλέον δυνατότητες για διάφορους ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένου και του κοινού, για να μπορεί να συμμετέχει και να εκφράζει την άποψή του στη διαδικασία λήψης απόψης. Παραδείγματος χάρη, ένα ελάχιστο ε, ε, χρονικό περιθώριο, ε, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή και όταν βλέπουμε και τι κάνουν τα κράτη-μέλη, θεωρήσαμε ότι εδώ δεν δινόταν επαρκής χρόνος στο κοινό και εμείς με την πρότασή μας θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι το κοινό θα έχει μια προθεσμία στη διάθεσή του προκειμένου να σχολιάσει και να συμμετέχει. Και μάλιστα με τρόπο ε, που θα τους επιτρέπει να εξετάζουν ενδελεχώς τις προτάσεις. Ωστόσο, κάποιες από τις τροπολογίες, και εδώ για παράδειγμα αναφέρομαι στην τροπολογία 22 για την δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία screening και υπάρχουν και κάποιες άλλες τροπολογίες που θέλουν να υπάρχει δημόσια συμμετοχή πριν ε, από την σύμφωνη γνώμη που θα πρέπει να δίνεται θεωρούμε ότι αυτό θα καθυστερήσει πάρα πολύ τη διαδικασία της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μάλιστα σε βαθμό που δεν θεωρούμε ότι θα μας διασφαλίζει ότι εφαρμόζουμε καλύτερα την περιβαλλοντική μας νομοθεσία και επίσης ε, θα μπορούσε να έχει και οικονομικές συνέπειες διότι μπορεί να οδηγεί σε καθυστερήσεις χωρίς λόγο. Όσον αφορά τις τροπολογίες για τα διορθωτικά μέτρα, τροπολογία 21 για παράδειγμα για την εκ των υστέρων παρακολούθηση έργων που έχουν πολύ σημαντικές αρνητικές συνήπειες, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε κατά την άποψή μας. Είμαστε θετικοί εν γέννη σε κάποιες από τις προτάσεις που γίνονται εδώ, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε και ότι δεν θα έχουμε και επιπλέον διοικητικό άχθος. Εδώ θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο συζήτησης. Να περάσω τώρα στην τρίτη κατηγορία τροπολογιών που θεωρώ ότι υπερβαίνουν ε, σαφέστατα τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτές δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε και θα ήθελα να σας συνοψίσω και τους λόγους ε, ακολουθώντας και το σχέδιο έκθεσης του εισηγητή. Για παράδειγμα, η πρόταση ε, τροπολογίας για τον ορισμό για τη βιοποικιλότητα, τροπολογία 13. Γνωρίζουμε ότι είναι περιττή αυτή η τροπολογία και για λόγους ε, νομικής απλούστευσης. Υπάρχει ένας πολύ σαφής ορισμός της βιοποικιλότητας ε, στη σύμβαση για την βιολογική ποικιλότητα στην οποία συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως η σύμβαση είναι τμήμα του κοινοτικού δικαίου και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον ορισμό όσον αφορά την τροπολογία η οποία επιτρέπει να ε, έχουμε παράταση στις χρονικές προθεσμίες μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εδώ θα ήθελα να σας παραπέμψω στα τη σύμβαση του Άρχους, η οποία προβλέπει ότι οι 45 μέρες επαρκούν. Η πρόταση έπρεπε να αφήσει αρκετή ευελιξία στα κράτη-μέλη και να δίνεται παράτηση ανάλογα με τη φύση, την πολυπλοκότητα και το μέγεθος του προτινόμενου έργου. Ελπίζω να συμφωνούμε όλοι ότι είναι τελείως διαφορετικό το ένα θέμα από το άλλο και το μέγεθο ενό έργου και το χρονοδιάγραμμα εντό του οποίο μπορεί να ληφθεί απόφαση. Αν έχουμε ένα πολύ περίπλοκο έργο ε, και είναι πολλά ε, τα στοιχεία, θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα παρέκκληση. Παρεπιπτόντω, θεωρούμε ότι πρέπει να είναι δεόντω αιτιολογημένο και η παράταση δεν είναι παόριστον, είναι μια παράταση η οποία δίνεται για ένα επιπλέον διάστημα τριών μηνών. Και πάλι λοιπόν είμαστε εντός των χρονικών ορίων ε, πολύ συγκεκριμένοι. Και τέλος, το σχέδιο έκθεσης αναφέρεται στο σχιστολιθικό φυσικό αέριο, το είπαν και πολλοί εδώ αρκετές φορές. Συμφωνούμε όλοι ότι το σχιστολιθικό φυσικό αέριο είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και το συζητούν όλοι, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απλώς συζητάται όλο ένα και περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πάρα πολλέ ιδιαιτερότητες το συγκεκριμένο ζήτημα και προτού λάβουμε οποιοδήποτε μέτρο, θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει ενδελεχή αξιολόγηση του ευρωπαϊκού πλαισίου, Γνωρίζετε ότι ο νομοθέτης ε, ε, και το, συγγνώμη, το νομοθετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής για το 2013 έχει συγκεκριμένες δράσεις όσον αφορά το σχιστολιθικό φυσικό αέριο και όταν προετοιμάσαμε και προτείναμε τη συγκεκριμένη αναθεώρηση της οδηγίας η αξιολόγηση ήταν εν εξελίξη ακόμα για το θέμα αυτό και επιπλέον οι δυνατότητες που έχουμε για τα παραρτήματα 1 και 2 θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση αντικτύπου για το θέμα του συστολιστικού φυσικού αερίου, γιατί είναι πάρα πολύ υψηλό το, το κόστος και θεωρήσαμε ότι δεν πρέπει να αναφέρομαστε συγκεκριμένα σε έργα συστολιστικού φυσικού αερίου. Και πρέπει βέβαια εδώ να πω ότι και τα έργα έρευνα και εξόρυξη χιστολιστικού φυσικού αερίου περιλαμβάνονται στο παράτημα 1 παρά το γεγονό ότι περιορίζονται ω προ τι ποσότητε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αξιολόγηση αντικτύπου που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα, ξανακάνουμε, τι θα κάνουμε με το θέμα αυτό. Ε, προτείνονται όμως και κάποιες ποιοτικέ αλλαγές, όπως για παράδειγμα την υποχρεωτική εξέταση εναλλακτικών λύσεων, παρακολούθηση, όλα αυτά ε, έχουν ε, ήδη σχέση με έργα σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Αν λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις συζητήσεις τους αναφερθούν περαιτέρω στο θέμα αυτό και έχουμε και εμείς περισσότερες πληροφορίες από πλευράς μας, τότε σαφώς είμαστε διατεθειμένοι να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα διότι είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον εισηγητή για την έκθεσή του και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοιχτή για να εξετάσει όλες τις τροπολογίες που στόχο έχουν να βελτιώσουν το σχέδιο κειμένου, ε, φυσικά το σκεπτικό και τους στόχους της πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τις παρεμβάσεις όλων των συναδέλφων τους, οποίους και ευχαριστώ για τις προτάσεις τους. Θα δούμε τώρα από τις προτάσεις αυτές ποιες ε, τροπολογίες θα προκύψουν Θα ήθελα να εκφράσω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια οδηγία η οποία επιβάλλει μια εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε έργα τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 1 τη στιγμή της εκτέλεσής τους μπορούν να διαρκέσουν ακόμα και 10 ή 20 χρόνια. Ορισμένα μάλιστα μπορούν να έχουν μια διάρκεια ζωή που διαρκεί και έναν αιώνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για πάρα πολύ σημαντικά έργα, τα οποία αποτελούν κληροδότημα και για τι επόμενε γενναίε. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, είναι λογικέ ανησυχίε οι οποίε έχουμε αυτή τη στιγμή σε σχέση με τι τοπικέ ε, εθνικέ αρχέ ή και σε σχέση με τον ε, κύριο του έργου όσον αφορά το κόστος, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Πιστεύω πάντως ότι το καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στα διάφορα στάδια της αξιολόγησης, ουσιαστικά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα κέρδος τόσο χρόνου πολλές φορές, ακόμα και οικονομικών όμως πόρων ή περιβαλλοντικών πόρων. Πολύ συχνά, καθώς προσπαθούμε πάρα πολύ γρήγορα να προχωρήσουμε μια διαδικασία, δεν καταφέρνουμε τελικά να συνειδητοποιήσουμε και ποια είναι η άποψη του διαφερόμενου κοινού και όταν είναι ενδιαφερόμενο κοινό, ουσιαστικά αναφέρομαι πολλέ φορέ ακόμα και στου Δήμου, τι μικρέ τοπικέ αρχέ. Αυτό το οποίο μα έχει διδάξει η πείρα είναι ότι πολλέ φορέ ο χρόνο που κερδίζουμε στην αρχή το χάνουμε στη συνέχεια μέσα σε αένεε νομικέ αντιπαραθέσει που έχουν διαρκέσει πάρα πολλέ φορέ πάρα πολλά χρόνια και σε ορισμένα κράτη-μέλη έχουν οδηγήσει και σε μπλοκάρισμα των έργων. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να μα απασχολήσει το ζήτημα αυτό, γιατί μιλάμε για πολύ σημαντικά έργα, ορισμένα εκ των οποίων είναι δημόσια έργα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια να καταφέρουμε να προστατεύσουμε στο πλαίσιο των έργων αυτών και τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογουμένου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών είναι 22 Μαΐου, 12 το μεσημέρι και θα εξετάσουμε πάλι τις τροπολογίες αυτές στις 19 και 20 Ιουνίου. Ιουλίου μάλλον και προβλέπεται, μάλλον Ιουνίου με συγχωρείτε και η ε, ψηφοφορία θα γίνει στις 10 Ιουλίου στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ για όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση και περνάμε στο σημείο 5. Εδώ θα δώσω αμέσως το λόγο στην συγγήτρια την κυρία Λεπάζου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα των βιοκαυσίμων είναι ένα θέμα ευαίσθητο, το οποίο θα έλεγα ότι πολλές φορές ε, προσκούει στη δυσκολία διαφορετικών και αντικρώμενων συμφερόντων. Οι ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας έχουν ε, τεθεί για το 2020 σαν στόχος με 20% σε γενικές γραμμές και 10% στις μεταφορές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτό το 10% για τις μεταφορές θα αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα γεωργικά καύσιμα. Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε σχέση με την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων. Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικά κείμενα τα οποία πρέπει να επεξεργαστούμε. Είμαι πολύ ευτυχής γιατί ο συνάδελφος Βιντάλ Κάντρας που είναι εισηγητής για την Επιτροπή Βιομηχανίας παρακολουθεί τις εργασίες μας και ξεκινάμε βέβαια από διαφορετικές ε, θέσεις, αλλά πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε μία κοινή θέση. Σκοπός όλων μας είναι να μειώσουμε τις εκπομπές ε, αερίων θερμοκηπίου. Το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει την ε, επιθυμία του να λάβουμε υπόψη μας όλους αυτούς τους παράγοντες που προκαλούν αλλαγές όσον αφορά την ποιότητα του εδάφους, αλλαγές και τροποποιήσεις που οφείλονται στην χρησιμοποίηση των αγροκαυσίμων. Είχαμε δώσει εντολή στην Επιτροπή να αναπτύξει μία μεθοδολογία που θα λάμβανε υπόψη της αυτόν τον παράγοντα. τον λεγόμενο παράγοντα Κάζι. Όσον αφορά λοιπόν τους διάφορους παράγοντες και τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν, μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε σε διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τις υποθέσεις εκκίνησης. Παρ' όλα αυτά όλοι διαπιστώνουν το φαινόμενο αυτό, το φαινόμενο Κάζι, η Ευρώπη δεν είναι η μόνη που έχει επεξεργαστεί αυτόν τον παράγοντα. Το ίδιο ακριβώ έχουν κάνει και οι Ηνωμένε Πολιτείε στα πλαίσια της ε, νομοθεσίας της Καλιφόρνιας, παραδείγματος χάρη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο παράγοντας Κάζι είναι πολύ πιο σημαντικός για τις πρώτες ύλε του βιοδίζελ σε σχέση με την παραγωγή εθανόλης, βιοεθανόλης. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε διαφανείς και ειλικρινείς, αν πραγματικά ο σκοπός μας είναι η μείωση των εκπομπών των αερίων ε, θερμοκηπίου, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον παράγοντα κάζι. Είναι απαραίτητο αυτό και κατά δεύτερο λόγο δεν μπορούμε και νομίζω ότι εδώ συμφωνούμε όλοι, να συνεχίσουμε μια πολιτική στην οποία πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ της διατροφής και των μεταφορών. Η επιλογή λοιπόν γεωργικής αγροτικής πρώτης ύλης για την δημιουργία καυσίμων οδηγεί σε αυτήν την ε, επιλογή. Σήμερα ο ειδικό συζητητής των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στην διατροφή, ο κύριος Ντεσούτερ, μας έχει στείλει ένα έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ο σημαντικός ρόλος όσον αφορά την κατανομή των ε, γεών, των εδαφών για την παραγωγή βιοκαυσίμων και αγροκαυσίμων. Βλέπετε ότι η πρώτη γενιά τέτοιων καυσίμων που παράγονται από γεωργικές πρωτεσίλες και που ουσιαστικά βασίζονται στην χρήση ε, φυτικών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την παραγωγή ειδών διατροφής είναι το αντικείμενο αυτής της πρώτης έκθεσης. Αν λάβουμε υπόψη μας λοιπόν τον παράγοντα Κάζη στον υπολογισμό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μπορούμε να ταξινομήσουμε σε καλές και κακές, αν θέλετε, παραγωγές σε σχέση με τον παράγοντα Κάζη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε κάποιες επιλογές όσον αφορά την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε χωρίς να ε, ορίσουμε έναν μοναδικό ενιαίο κανόνα ο οποίος θα ισχύει παντού κάτι που είναι δύσκολο να γίνει κατά την απόψή μου. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις μέχρι τώρα επενδύσεις που έχουν γίνει πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τη μείωση βεβαίως των εκπομπών του αεροθερμοκηπίου αλλά και μια παγκόσμια λογική σε σχέση με την παραγωγή ειδών την οικονομική κρίση και δεν είναι δυνατόν κάποιος να αγνοήσει το γεγονός ε, ότι οι αποφάσεις που παίρνουμε έχουν επιπτώσεις ε, στη βιομηχανία. Γι' αυτό και στην έκθεσή μου σας έχω προτείνει να εφαρμόσετε την ε, ρήτρα grandfather όσον αφορά την παραγωγή καυσίμων από ε, γεωργικές πρωτεσίλες της πρώτης γενιάς και να ξαναδούμε βεβαίως ε, τις ε, ε, ημερομηνίες όπως τις είχαμε καθορίσει ξεκινώντας από το 2010. 4,3% επί αυτού του 10% για το ε, βιολογικό ντίζελ. Όσον αφορά την εθανόλη, εδώ ο παράγοντας δεν είναι καλός, όπως είπαμε, η ταξινόμηση δεν είναι καλή, θα πρέπει λοιπόν όσον αφορά την εθανόλη να μην ξεπεράσουμε το 2,25% για το 2020. Ε, Αυτό προτείνει η Επιτροπή. Και για να φτάσουμε μέχρι το 2020, εγώ σας προτείνω να καταργηθούν οι επιδοτήσεις για τα καύσιμα αυτά τα οποία δεν έχουν θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στο κλίμα και η στήριξη, αν θέλετε, σε αυτόν τον τομέα, όπως ξέρουμε, είναι πολύ σημαντική. Είναι περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στα πλαίσια των δημοσιονομικών περικοπών που γνωρίζουμε στην Ευρώπη. Σας κάνω λοιπόν μια ισορροπημένη πρόταση. Ναι, μείωση αν θέλετε αυτών των καυσίμων πρώτης γενιάς που έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Ναι, να ενισχύσουμε τις επενδύσεις που έχουν γίνει μέχρι τότε ώστε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι αν θέλετε ένα ισορροπημένο σύστημα που σας προτείνω. Παρ' όλα αυτά, σκοπός μας είναι να φτάσουμε στο στόχο μας που είναι αυτό το 10%. Αν προσθέσω 4,5 και 2,25% απέχω από το 10%. Σας προτείνω λοιπόν έναν ε, στόχο μεσοπρόθεσμο, αν θέλετε, μέχρι το 10%. 1,5% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις μεταφορές. Προσθέτουμε λοιπόν αυτό το 1,5% και φτάνουμε στο 8%. Αυτό το 2% λοιπόν, όπως προτείνει ο κύριος Βιντάλ Κάντρας, θα καλυφθεί από αυτά τα δύο καύσιμα δεύτερης γενιάς, όπως το ονομάζουμε. Εδώ πρόκειται για μια λύση πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε κάποια υποπροϊόντα, θα έλεγα, διαφόρων τομέων και δραστηριοτήτων. Πρόκειται όμως για μια επιλογή η οποία αντιμετωπίζει, ε, προσκρούει μάλλον σε κάποιες δυσκολίες. Κάποιες από αυτές τις προτάσεις ήδη χρησιμοποιούνται, παραδείγματος χάρη Κάποια από τα ζωικά λύπη χρησιμοποιούνται ήδη στη χημεία. Κάποια προϊόντα ξυλίας που χρησιμοποιούνται ήδη για την παραγωγή χαρτιού. Είναι λοιπόν πολύ συγκεκριμένη, αν θέλετε, η επίπτωση, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχουν εδώ κοινωνικές συνέπειες, οικονομικές συνέπειες, ε, θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε κάποιες ε, αποφάσεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε κάποιες βιώσιμες επιλογές. Δεν θα πρέπει σε λίγα χρόνια εμείς ή αυτοί που θα ακολουθήσουν στη θέση μας να αναγκαστούν να πούν ότι κάναμε λάθος. Οι αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα έχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις όσον αφορά αυτά τα βιοκαύσιμα και θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση των συνεπειών και των επιπτώσεων και από οικονομικής και από κοινωνικής απόψεως, έτσι ώστε να μην αποσταθεροποιήσουμε οικονομικές δραστηριότητες που υπάρχουν και λειτουργούν ικανοποιητικά. Αυτά όσον αφορά τα βιοκαύσιμα δεύτερης ή τρίτης γενιάς με τα φύκια. Και τελειώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στην ξυλία στη δασοκομεία. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ένας τομέας εξαιρετικά σημαντικός για την Ευρώπη. Ίσως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Γι' αυτό και στην έκθεσή μου σας προτείνω να μην ε, ενθαρρύνουμε την χρήση στα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς προϊόντων ξυλίας. Και αν το κάνουμε θα πρέπει προηγουμένως να διαπιστώσουμε ότι η ανάπτυξη των δασών μας επιτρέπει κάτι τέτοιο. Σήμερα έχουμε την ξυλία για την παραγωγή ενέργειας, για την παραγωγή χαρτιού και για τα βιοκαύσιμα. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να σιγουρευτούμε ότι δεν καταστρέφουμε τα δάση μας για να τα εκμεταλλευτούμε σε όλους αυτούς τους τομείς. Προτείνω λοιπόν εδώ να υπάρχει μία ρήτρα βιωσιμότητας όσον αφορά τουλάχιστον τη χρησιμοποίηση των προϊόντων ε, ξυλίας για τα βιοκάψιμα δεύτερης και τρίτης γενιάς. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η πρότασή μου είναι ισορροπημένη. Άκουσα πολλές απόψεις, πολλούς παρεμβαίνοντες. Σκοπός μας είναι η μείωση των εκπομπών ε, αερίου θερμοκηπίου. Ελπίζω η πρόταση να είναι βιώσιμη και με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσω τις παρατηρήσεις ε, όλων σας. Merci. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Βίλα Κβάντρας από την Επιτροπή Βιομηχανίας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας που μου δίνετε τη δυνατότητα να συμμετέχω και εγώ στις ε, συζητήσεις σας εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή για μένα που είμαι μέλος Επιτροπής Βιομηχανίας να φτάνω εδώ πέρα στην ε, καταπληκτική αυτή επιτροπή που τόσο στεναρά προστατεύει, την προστατεύει το περιβάλλον. Θα ήθελα με ιδιαίτερη μετριοπάθεια να ανταποκριθώ στα όσα μας είπε η κυρία Λεπάζ, καθότι γνωρίζουμε ήδη το περιεχόμενο της έκθεσής της, την οποία παρουσίασε και στη δική μας την Επιτροπή και είχαμε ήδη δυνατότητα να κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων μαζί της. Συμφωνώ με την κυρία Λεπάζ ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο από οικονομική, κοινωνική και τεχνική πλευρά. Συνεπώς υπάρχουν πολλά επιμέρου στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και βέβαια πολλές διαφορετικές ε, προσεγγίσεις που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε, οι οποίες είναι απόλυτα νόμιμες και λογικές. Ο συνήθως όμως εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε έναν κοινό τόπο, μια κοινή κατεύθυνση, ένα σημείο σύγκλησης όπου θα καταφέρουμε τελικά να συγκεράσουμε όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις, συμφέροντα και στόχους. Είμαι πεπισμένος ότι οι δυο μας επιτροπές θα καταφέρουν να συνεργαστούν με απόλυτη ειλικρίνεια και επικοδομητικά προς τον στόχο αυτό και θα καταφέρουμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της έμεσης αλλαγής της χρήσης γης. Εγώ είμαι στην απόλυτη διαθεσιμότητά σας. Στη δική μου την Επιτροπή σήμερα είναι η καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Πολύ σύντομα λοιπόν θα είμαι σε θέση να έχω μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της τελικής γνωμοδότησης και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω τότε τη συνεργασία και την ειδική σα την Επιτροπή. Τώρα, όπω και η κυρία Λεπά, θα ήθελα και εγώ πολύ σύντομα να σα παρουσιάσω τη δική μου προσωπική άποψη, εφόσον είμαι συντάκτη γνωμοδότησης, όπω το καταλάβατε, για το ζήτημα αυτό στην Επιτροπή ε, βιομηχανία. Καταρχά να αναφερθώ στον στόχο της μείωσης του φαινομένου ILUC, του φαινομένου της έμεσης αναλλαγής της χρήσης γης. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινό στόχο όλων μα. Εφτά είναι οι επιτροπέ οι οποίε ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, με το υποεξέταση νομοθέτημα, εκ των οποίων οι έξι έχουν ήδη υποβάλει την πρότασή του και με την εξαίρεση της έκθεσης κυρίας Λεπάς, κανεί δεν είναι υπέρ τη συμπεριληψη του συντελεστή ILUC με δεσμευτικό τρόπο στην έκθεση αυτή. Καταλαβαίνετε ότι το στοιχείο αυτό έχει μία ποσοτική πλέον διάσταση και νομίζω ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αναθεώρηση και την εξέταση διαφόρων μελετών και έχοντας κάνει και η ίδια τη δική της την έρευνα, γνωρίζει πλέον πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά επιστημονικά δεδομένα προκειμένου να μπορούμε με βεβαιότητα να βάλουμε συγκεκριμένες οριακές τιμές για κάθε είδος προϊόντος για κάθε φυτή, φυτικό προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται. Ξέρετε ότι στη δική μου τουλάχιστον επιτροπή υπάρχουν ορισμένα άτομα τα οποία έχουν σημαντικές επιστημονικές σπουδές διατελέσει στο παρελθόν. Επομένως γνωρίζουν ότι ορισμένα στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν τμήμα ενός συγκεκριμένου μοντέλου. Θεωρώ ότι Πέρα από τη μοντελοποίηση αυτή, εμεί θα πρέπει να δώσουμε μια απαραίτητη ασφάλεια δικαίου και βεβαιότητα στι παραμέτρου οποίε εξετάζουμε και πεντάσουμε στην έκθεση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βαζόμαστε μόνο σε πράγματα τα οποία μπορούμε να υπολογίσουμε. Το να ενσωματώσουμε τώρα στο νομοθέτημα αυτό κάτι το οποίο μπορούμε μόνο να μοντελοποιήσουμε στη φάση αυτή, για το οποίο μπορούμε να καταρτήσουμε δηλαδή μόνο μοντέλο, είναι κάτι το κάπως επικίνδυνο θα έλεγα. Χρησιμοποίησα και εγώ μία έκθεση την οποία χρησιμοποίησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταφέρουμε να ποσοτικοποιήσουμε τον παράγοντα ILUC και η μελέτη αυτή όντως αναφέρεται σε συγκεκριμένες αδυναμίες και βεβαιότητα όσον αφορά τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ότι η Μαλαισία, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγούς τέτοιων καυσίμων, Φανταστείτε λοιπόν ότι η Μαλαισία εγκρίνει κάποια στιγμή στο μέλλον ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα το οποίο θα απαγορεύσει την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων. Χρησιμοποιώντας, καταλαβαίνετε ότι για το, για το φινικέλαιο πρόκειται να τροποποιηθεί εντελώς ο συντελεστής άελουκ ο οποίος χρησιμοποιείται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με παράγοντες οποίους δεν ελέγχουμε εντελώ, με συντελεστές στους οποίους δεν ορίζουμε εντελώ. Επίσης ο συντελεστής ILUC χρησιμοποιείται πολλές φορές προκειμένου να γίνεται μια διάκριση ανάμεσα στην εθανόλη και το βιοντίζελ. Αν χρησιμοποιηθεί όμως ο συντελεστής αυτός, τότε θα πρέπει να δούμε και τι συνέπειες θα μπορεί να έχει μετά την εφαρμογή του και πολύ φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε στο ακόλουθο σενάριο. Θα έχουμε πλήρη εξαφάνιση του βιοντίζελ, ενώ η εθανόλη που αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ χαμηλό συντελεστή αελουκ, θα έχει έναν τέτοιο συντελεστή αελουκ υψηλότερο στο μέλλον, ο οποίος ήταν τελικά επιζήμιος για την εθανόλη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε πολύ επικίνδυνα νερά και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχουμε λοιπόν το στόχο του 10% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2020 στον τομέα των μεταφορών. Πρέπει να επιτύχουμε το στόχο αυτό σίγουρα. Αλλά ας επιλέξουμε σωστά τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουμε το στόχο αυτό. Όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος. Αλλά ας ακολουθήσουμε τουλάχιστον την καλύτερη δυνατή μέθοδο. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε έχουμε και αυτή τη συζήτηση τώρα. Θεωρώ ότι μια επικοδομητική προσέγγιση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη και πολλές, πολλά διαφορετικά πλεονεκτήματα τα οποία έχουν τα βιοκαύσιμα, γιατί έχουν πλεονεκτήματα όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την ανεξαρτησία της ενέργειας και την ανάπτυξη της υπαίθρου, μπορεί να εγκριθεί λοιπόν με τέτοια προσέγγιση, προκειμένου να καταφέρουμε να μειώσουμε το φαινόμενο της έμεσης αλλαγής της χρήσης γης. Οι περισσότεροι άλλωστε συμφωνούν ότι τα προηγμένα βιοκαύσιμα έχουν πλεονεκτήματα, και ξέρω ότι τα βιοκαύσιμα αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση, δεν βάλουν κατά τι καλλιέργειε και τη παραγωγή τροφίμων. Α τα προωθήσουμε λοιπόν, αλλά πώ θα το κάνουμε αυτό. Η κύριε Λεπάζα έχει απόλυτο δίκιο. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο αν θέσουμε ένα συγκεκριμένο υποστόχο για τα βιοκαύσιμα, για τα προηγμένα βιοκαύσιμα. Μπορούμε να έχουμε ένα επιμέρο, επιμέρους στόχο για τα βιοκαύσιμα αυτά, τα οποία μπορεί να είναι 5% για παράδειγμα, και κατά αυτόν τον τρόπο θα στείλουμε προς τις αγορές και προς το βιομηχανικό κλάδο ένα συγκεκριμένο μήνυμα, όπως άλλωστε κάναμε το 2009 με το στόχο του 10%. Και αυτή τη φορά θα στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, το οποίο θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις στα προηγμένα βιοκαύσιμα. Συμφωνούμε νομίζω όλοι στο σημείο αυτό, να έχουμε έναν επιμέρους στόχο για τα προηγμένα βιοκαύσιμα. Ο στόχος αυτός τώρα μπορεί να συμπληρωθεί μέτρα μείωσης της έμεση αλλαγής της χρήση γης, όπως άλλωστε έχει εξηγηθεί σε πάρα πολλές ε, εκθέσεις που έχουν ε, υποβάλει η WWF, διεθνείς ε, φορείς ή το Πολυτεχνείο της Λοζάνης ή άλλοι οργανισμοί, οι οποίοι είναι οργανισμοί ιδιαίτερης έγκλης κιόλας. Στόχος πάντως είναι να ενθαρρύνουμε τις πρώτες ύλε εκείνες οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των καυσίμων αυτών. Καταλαβαίνετε ότι χρησιμοποιώντα τι πρώτε αυτέ ύλε μειώνεται το φαινόμενο τη έμεση αλλαγή τη χρήση γη και δεν υπάρχει καμία στρέβλωση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, την αγορά και την απασχόληση. Μια τελευταία παρατήρηση. Πρέπει να σα πω ότι δεν έχουμε ακόμα πολλέ πράσινε εναλλακτικέ λύσει για να αντικαταστήσουμε τα βιοκαύσιμα. Όπως θα έχετε καταλάβει, σε καμία περίπτωση δεν είμαι κατά. Αντίθετα, είμαι σαφώς υπέρ της χρησιμοποίησης ηλεκτρικής ενέργειας της μεταφορές. Νομίζω ότι θα πρέπει όλο και περισσότερο να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτή στο μέλλον και να έχουμε όλο και πιο αποτελεσματικές, αποτελεσματικούς κινητήρες αν θέλετε. Οι επενδύσεις όμως αυτές δεν αρκούν για να καλύψουμε το κενό το οποίο θα παρουσιαστεί μέχρι το 2020. Άρα έχουμε το ακόλουθο δίλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δίλημα το οποίο είναι δυσυπήλυτο σίγουρα. Είτε θα εγκαταλείψουμε το στόχο του 10% για τις νόμιμες πηγές ενέργειας στον τομέα των μεταφορών και νομίζω ότι η πολλαπλή προσμέτρηση ουσιαστικά, είναι ένας, ουσιαστικά σε αυτό αντιστοιχεί μέσω της πολλαπλής προσμέτρησης, ουσιαστικά τι λέμε. Λέμε ότι εγκαταλείπουμε το στόχο του 10%. Ας μην γελιόμαστε. Μπορούμε να το συγκαλύψουμε με διάφορους τρόπους, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και πρέπει μεταξύ μόνο τουλάχιστον να είμαστε ειλικρινείς. Κύριε Πρόεδρε, με την άδειά σα να αναφερθώ και σε μια πρόσφατη εμπειρία που είχα. Τι τελευταίε αυτέ εβδομάδε, πέντε μέλη πήγαμε στην Μαλαισία σε μια διαβεντική αποστολή όσον αφορά το φινικέλαιο. Μιλήσαμε με τι αρμόδιε αρχέ τη χώρα αυτή, μιλήσαμε με εκπροσώπου βιομηχανίας, με εκπροσώπου μη κυβερνητικών οργανώσεων, με εκπροσώπους ναυτοχθόνων, με του πάντες μιλήσαμε. Και από ό,τι φαίνεται όλοι συμφωνούν ότι θέλουν το φινικέλαιο να χρησιμοποιηθεί ως βασικό στοιχείο της οικονομίας τους. Ολοκληρώσει παρακαλώ πολύ ο Πρόεδρος. Ναι. Αυτό το οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε όμως είναι οι φοιτίες αυτές να επιτευχθούν χωρίς όμως να έχουμε αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και νομίζω ότι συμφωνούμε και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το στόχο αυτό. Συνοψίζοντας λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι να πω τα ακόλουθα. Χρειαζόμαστε έναν επιμέρου στόχο για τα προηγμένα βιοκάψιμα. Ε, χρειαζόμαστε θετικές επιπτώσεις μείωσης του ILUC και θα πρέπει μέσω της δικής μας εμπορικής πολιτικής να προωθήσουμε δεσμευτικά μέτρα τα οποία να ισχύουν για όλους τους διεθνούς μας εταίρους. Νομίζω ότι αυτή είναι τουλάχιστον αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε και αυτόν προτείνω εγώ ως συντάκτης νομοδότης στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Δακάντρας. Για μας είναι σπάνιο και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συναδέλφους από την Ήτρε. Είναι τεράστιο το θέμα, είναι πολύπλοκο και σίγουρα θα πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί έτσι ώστε να προχωρήσουμε όλοι προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι σκιώδεις εισηγητές και οι υπόλοιποι ομιλητές. Τέσσερα λεπτά για τους σκιώδεις έχουμε, κατόπιν Αγιούζο, Πέτερ Χάιμας, Σέμπερ. Ποιος άλλος έχει ζητήσει το λόγο, Ήβκοσε. και κυρία Γκάρλινγκ. Να ξεκινήσουμε όμως με τους σκιώδεις εισηγητές. Η κυρία Κλάς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα και βλέπετε ότι και η συζήτηση αυτή συμπεριλαμβάνει πολλά θέματα. Ακούσαμε την εισηγήτρια την κυρία Λεπάζ, η οποία έθεσε πολλά θέματα, το ίδιο έκανε και ο συνάδελφο από την Επιτροπή Ήτρε. Νομίζω ότι όταν ξεκινήσαμε με τους στόχους, ήμασταν πολύ ενθουσιώδεις, θέσαμε τους στόχους μα 10%, ήταν ένας στόχος πραγματικά ο οποίος μας οδήγησε σε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και στον ε, κανονισμό. Διαβάζοντας όμως την έκθεση της Κορίν Λεπά συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να ξαναδούμε κάποιους στόχους. Είναι αυτή η βιώσιμη πολιτική. Γιατί πρέπει να δούμε πολύ συγκεκριμένα τα στοιχεία και τα πραγματικά γεγονότα. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε ούτε να τα παρεκκλίνουμε. Γι' αυτό και θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε για τα επόμενα χρόνια για τις μεταφορές, την ενέργεια με παραδοσιακούς τρόπους ε, και παραδοσιακά καύσιμα. Βεβαίως σκοπός μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Βεβαίως σκοπός μας είναι να αυξηθεί η αηφορία. Βεβαίως και πρέπει να δούμε το θέμα της ενέργειας, η έλλειψη ανεξαρτησίας ε, όσον αφορά την ενέργεια κάτι που χαρακτηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε όταν παίρνουμε αυτές τις αποφάσεις. Και γι' αυτό και σήμερα μιλούμε για την έμεση αλλαγή στη χρήση γης. Αυτό βάσει πολύ συγκεκριμένων κριτηρίων που όπως μας είπε και ο συνάδελφος Βιντάλχαδα από την Επιτροπή Ιτρέ δεν είναι ένας επιστημονικός και απόλυτα ακριβής τρόπος μέτρησης. Έχουμε σήμερα δει ότι πολλές ε, αδυναμίες του συστήματος οφείλονται σε ανακριβείς υπολογισμούς. Και αυτό το έχει ε, αναγνωρίσει η Επιτροπή και το γνωρίζει πολύ καλά και η Κορίν Λεπάζ. Σήμερα λοιπόν έχουμε τους συνταλεστές ε, αυτούς οι οποίοι υπολογίζουν πολύ συγκεκριμένα τις εκπομπές την ε, παραγωγή αερίων, την συμβολή των τροπικών δασών και την πιστοχώρηση κάποιων εκτάσεων, την μείωση συγκεκριμένων εκτάσεων, κάτι που συμβαίνει καθημερινά. Τα δεδομένα που έχουμε όμως πρέπει να είναι πραγματικά ενημερωμένα, επίκαιρα. Και βλέπουμε ότι σήμερα ο συντελεστής της έμεσης αλλαγής για τη χρήση γης δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν αμετάβλητος και απόλυτα ακριβής. Και αυτό επαναλαμβάνω το αναγνωρίζει η Επιτροπή, κάτι που σημαίνει ότι μία βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να βασίζεται σε πολλούς συντελεστές και όχι σε έναν μοναδικό, κυρίως όταν αυτός εμπεριέχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα και ασάφεια. Χρειάζονται επενδύσεις στην καινοτομία. Ναι, αυτό όμως καταλαβαίνετε ότι μπορεί να βασίζεται μόνο σε μια ασφάλεια αυτών των επενδύσεων. Η Κορίνη Λεπάζ αναφέρεται επίσης στο grandfathering, λέγοντας ότι αυτό μας δίνει περισσότερη βεβαιότητα. Τι να σας πω, κοιτάξτε τις ε, προοπτικές επενδύσεων και βάσει αυτών θα πρέπει να στηρίξουμε τις μελλοντικές πολιτικές μας αποφάσεις οι έρευνες που βασίζονται στο συντελεστή έμεσης αλλαγής της χρήσης γης μας δίνουν σήμερα ένα σημαντικό ποσοστό αβεβαιότητας. Βεβαίως η ευρωπαϊκή παραγωγή θα πρέπει να δώσει κίνητρα στην βιώσιμη ανάπτυξη, στη βιώσιμη ε, παραγωγή και βλέπετε ότι εδώ ακόμα και αν δούμε τα στοιχεία των ε, μη κυβερνητικών οργανισμών η βιωσιμότητα της παραγωγής, ένα καθαρό περιβάλλον, ζητά από όλους εμάς, εμάς τους Ευρωπαίους, μία πιο σαφή ρύθμιση. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε όμως αυτή την αηφορία, αυτή τη βιωσιμότητα. Έχουμε θέσει ένα στόχο, 10%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ μας προτείνει αυτό το 5%. Δεν δεχόμαστε τέτοιου είδους μη δικαιολογημένε μειώσεις και πιστεύω πραγματικά ότι όσον αφορά το ποσοστό 40%, 60%, το μείγμα των ουσιών και των πρώτων υλών. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε παραδείγματο χάρη τα βιοκαύσιμα και τα απορρίμματα. Με συγχωρείτε πρέπει να διακόψετε. Έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας κατά 1,5 λεπτό. Κοιτάξτε, έχουμε μια ομερήσια διάταξη. Δεν μας επιτρέπει ο χρόνος. Ο Κρίδων Αρσέντσιθο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Σποκ θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω. Ο κύριος Αρσένης θα ήθελε να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την εξαιρετική προσέγγιση που ακολούθησε στο θέμα αυτό η πολιτική σας βοηθά τα βιοκαύσιμα και την επίτευξη του στόχου της μείωσης κατά 10% ε, των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών και μας ενδιαφέρει η κατάλληλη χρήση των βιοκαυσίμων. Ο στόχος είναι να μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου ως τμήμα της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος και φυσικά θα πρέπει να βοηθήσουμε με την ε, ε, κατάλληλη στήριξη για τα κατάλληλη χρήση των βιοκαυσίμων στα περισσότερα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η επίπτωση των βιοκαυσίμων αυτών είναι όντως ε, σημαντική. Δυστυχώς όμως τα κριτήρια εφορίας προς το παρόν ε, παραβλέπουν κάποιους παράγοντες, κυρίως για την έμεση αλλαγή χρήσης γης το επιστημονικό έργο καταδεικνύει ότι οι εκπομπές από την έμεση αλλαγή της ε, χρήσης γης μπορούν να μειώσουν ε, ποσοστό ή και όλα τα ωφέλη που έχουμε από την ε, χρήση βιοκαυσίμων. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης αυτής για την οδηγία είναι ο συνυπολογισμός της συνεισφοράς των βιοκαυσίμων και των βιοραυστών από τρόφιμα και ζωοτροφές. Ο κύριο Αρσένη συμφωνεί απόλυτα με το στόχο του ανώτατου αριού του 5% που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρεί ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πρότασης. Ο κύριος Αρσένης επίσης συμφωνεί με την πρόταση του εισηγητή να υπάρχουν ε, υποχρεωτικοί συντελεστές ε, iLook ε, και θεωρεί ότι το ποσοστό το οποίο αφορά τις μεταφορές δεν αποδίδει σωστά τους συντελεστές έμεσης αλλαγής της χρήσης γης και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να λάβουμε κατάλληλα μέτρα ώστε να έχουμε το στόχο του 30% από ανάσχημες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε περισσότερο περισσότερες ε, βιοκαύσιμα από τρόφιμα και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερα καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να επιτύχουμε το στόχο που θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κερδίσαμε λίγο χρόνο, χάρη σε εσάς. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο των τεσσάρων λεπτών. Δεν είναι όμω εύκολο για κάτι τόσο σημαντικό. Καταρχά, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Λεπάζ, για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και για την έκθεσή τη, η οποία αναφέρεται σε όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά και τον κύριο Βιντάλ Κουάντρα για τα όσα μα είπε εν είδη εισαγωγής. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι το ζήτημα του Άιλουκ δεν είναι καινούριο ζήτημα. Ήδη το 2008, όταν συμφωνήσαμε για το πακέτο κλιματικής αλλαγής, το κοινοβούλιο ήταν αυτό το οποίο ζήτησε να υπάρχουν συγκεκριμένα κρατήρια τα οποία να λαμβάνουν υπόψη του στην έμεση αλλαγή της χρήσης γης. 2008. Και βέβαια, δυστυχώ, χρειάστηκε να εγκαταλείψουμε τη θέση μα αυτή σε πραγματεύσει που είχαμε το Συμβούλιο. Και αυτό που λάβαμε ω αντάλλαγμα ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επέβαλε μια νέα έκθεση για το αν τελικά θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο συντελεστή ILUC ή όχι. Και βρισκόμαστε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Κάτι το οποίο ζητήσαμε εμεί στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο παρελθόν. Ανταποκρίνεται τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όχι πλήρω όπω θα έπρεπε για το ILUC. Γιατί καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ILUC είναι πρόβλημα και εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι δεν υπάρχει κανένας επιστήμονας αυτή τη στιγμή ο οποίος να λέει ότι δεν υπάρχει έμεση αλλαγή της χρήσης γης εξαιτία των βιοκαυσίμων. Το θέμα είναι πώς μπορούμε όμως να διευθετήσουμε το ζήτημα αυτό στα πλαίσια ενός νομοθετήματος. Αν εμείς καταλήξουμε στο να μην χρησιμοποιήσουμε συντελεστή ILUC, ουσιαστικά δίνουμε στο στελεστή αυτόν μηδενική αξία. Οτιδήποτε και να κάνουμε, δίνουμε τελικά μία τιμή, λαμβάνουμε μία απόφαση για το ILUC. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε να λάβουμε μία απόφαση για το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι θα κάνουμε εμεί με το ILUC. Θα ακολουθήσουμε τη γνώμη των επιστημών θα τους λα... ή όχι. Ζητήσαμε εμείς να υπάρξουν κάποια μοντέλα, μοντέλα τα οποία διεξάγονται, αυτή τη στιγμή βελτιώνονται, πολλές φορές να δεχομένως να μην λαμβάνουν υπόψη τους τα, παρα, τα παραπροϊόντα, τα μοντέλα αυτά, αλλά ήδη και τα μοντέλα αυτά ουσιαστικά έχουν ε, βελτιωθεί, εξελίσσονται σε καθημερινή βάση και προς τον κύριο Βιντάλ Κουάντρας να πω το εξή. Μα είπε ότι θα πρέπει να βασίζουμε την πολιτική μα σε μοντέλα. Εγώ θα έλεγα πηγαίνετε στον κύριο Λιρέν, ο οποίο βασίζει ουσιαστικά την πολιτική του λιτότητα σε καθημερινή βάση, βάση οικονομικών προβλέψεων, εκτιμήσεων και βασίζεται σε οικονομικά μοντέλα τη τάξη του 3%. Κάθε μέρα αυτό κάνει ο κύριο Ολιρέν. Εκτό μικροφώνη απάντηση. Ναι, αλλά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τον υποστηρίζει μέχρι στιγμή αν καταλήξουμε στο συμπέρασμα τελικά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τάστε κατά της λιτότητας, τότε και αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα για σήμερα. Πάντως, τα περισσότερα μοντέλα δείχνουν τελικά ότι όσο μεγαλύτερη η ύφεση, τόσο, πιο δυνάνει και τα αποτελέσματα τελικά. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα των συγκεκριμένων καταποκοπήν τιμών, δεν ξέρω αν μπορούμε πραγματικά να αποκλίνουμε. Ήδη υπάρχει μια οδηγία η οποία προβλέπει διατάξει για το ζήτημα αυτό. Όσον αφορά τώρα τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, αν μπορεί να δείξει κανεί ότι έχει τελικά χαμηλότερες τιμές, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις χαμηλότερες αυτές τιμές. Για ποιο λόγο να μην χρησιμοποιήσουμε τη διάταξη αυτή και για την έμεση αλλαγή της χρήση γη. Επομένως, είναι περίεργο ότι ξαφνικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστοχωρεί στο αν τελικά θέλει να κάνει κάτι με την έμεση αλλαγή της χρήσης γης. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να δούμε πώς θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τα προηγμένα βιοκαύσιμα, τα οποία ανταγωνίζονται λιγότερο την παραγωγή τροφίμων. Ο ανταγωνισμός αυτός υπάρχει. Τι μπορούμε λοιπόν εμείς να κάνουμε για τα προηγμένα βιοκαύσιμα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βεβαιότητα στους επενδυτές, ότι όσο πιο προηγμένα είναι τα βιοκαύσιμα, ε, τόσο πιο θετικές και επενδύσεις τελικά. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα στόχο και να σκεφτούμε και λίγο πιο πέρα από το 2020, δηλαδή να καταρτήσουμε μια στρατηγική που θα μας οδηγήσει πιο μακριά στο μέλλον. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους στόχους, όχι τεχνολογικούς αυτή τη στιγμή, αλλά στόχους οι οποίοι θα ξεπερνάνε ακόμα και το 3% για την περίοδο μετά το 2020. Πρέπει να καταφέρουμε μέσω των στόχων αυτών να μειώσουμε τους, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να περάσουμε πέρα από το 2020 όπως μας είπε και η κυρία Λεπάζ, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε για το ποσοστό 6% μέχρι το 2020 και να πάμε στο 10% για την περίοδο 2020 και μετά. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα θέτουμε στόχου για μια συγκεκριμένη τεχνολογία, αλλά θα θέτουμε στόχου για τη μείωση νερού θερμοκηπίου. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι στόχοι μα έχουν να κάνουν με συγκεκριμένε τεχνολογίε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω και είναι περίπλοκο το ζήτημα, η κυρία Γκίρλινγκ. Και είναι πολύ δύσκολο να επιτύχουμε πολλά πράγματα με τη μία. Και Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δεχτούμε ότι εξετάζουμε ρυθμίσεις στον κανονισμό επειδή υπάρχουν προβλήματα στον προηγούμενο κανονισμό και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Οι βασικές μας αρχές πρέπει να είναι απλούστευση, να μην είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα, να υπάρχει συνέπεια και σαφήνεια κυρίως για τις επενδύσεις και ίσω να υπάρχει και μια κάποια ευελιξία και να αναγνωρίσουμε το γεγονό ότι δεν είναι πολύ σαφεί οι επιστημονικές ενδείξεις όπως θα θέλαμε ε, και ίσω θα πρέπει να κάνουμε αλλαγέ ε, στην πορεία. Υπάρχουν πολλά και διάφορα θέματα τα οποία μα απασχολούν και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εξετάζουμε το καθένα μεμονωμένα, διότι όλα είναι και αλληλένδετα και όλα συνθέτουν ένα πάζολ. Και επομένω, είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε ε, τις ε, σαφείς, ε, ξεκάθαρες επιπτώσεις της ε, πρότασης της κυρίας Λεπάζ. Αντί λοιπόν να τα κοιτάω ένα-ένα αυτά, θα σας δώσω κάποιες συνολικές σκέψεις. Ο λόγος για τον οποίο κάνουμε τις νομοθετικές αλλαγές υποτίθεται ότι είναι ότι η αλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα στα βιοκαύσιμα δεν αυξάνει ε, τις ε, εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου μέσω της άμεσης αλλαγής της χρήσης γης και θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει αυτή η, η αύξηση πριν κάνουμε τις αλλαγές και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει επιστημονική βάση και κατάλληλη μεθοδολογία για να καθορίσουμε το κατάλληλο συντελεστή άϊκλου. Συμφωνώ ότι έγιναν κάποιε βελτιώσει, αλλά δεν είμαι απόλυτα βέβαιη ότι έχουμε επιτύχει το στόχο, όπω είναι ο κ. Βιντάλ Κρακουάντρας. Και δεν νομίζω ότι ο συντελεστή αυτό μα δίνει τι απαντήσει. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα προηγμένα βιοκαύσιμα. Δεν θα πρέπει να βασιστούμε απόλυτα σε κάτι το οποίο δεν υπάρχει ακόμα. Ξέρω ότι είναι καθοδόν, αλλά ε, και βεβαίω όλοι θεωρούμε ότι αν δώσουμε κίνητρα για επενδύσει θα έχουμε προηγμένα βιοκαύσιμα. Ωραία, στο ελπίσουμε, αλλά μην το θεωρήσουμε δεδομένο. Δεν μπορεί να είναι απαραίτητα τόσο εύκολο όσο νομίζουμε. Τώρα, όσον αφορά το ανώτατο όριο, και το ερώτημα για το κατά πόσον αυτό είναι το σωστό επίπεδο. Δέχομαι την αρχή ενό ανώτατου ορίου, αλλά δεν ξέρω αν το 5% είναι το κατάλληλο όριο. Κάποιε χώρε ήδη το έχουν υπερβεί και δεν ξέρω κατά πόσον ε, αφορά ε, μόνο συγκεκριμένο τομέα. Ίσως θα μπορούσαμε να το έχουμε και σε άλλους τομείς ε, και να έχουμε αυτή τη σωστή μεθοδολογία. Όσον αφορά τώρα την πολλαπλή προσμέτρηση, νομίζω ότι είναι επικίνδυνη. Και πάλι καταρχήν μια χαρά είναι, αλλά δεν υπάρχει κατάλληλη αξιολόγηση των επιπτώσεων και η λογική των δύο καταλόγων θα ήθελα πραγματικά να την εξετάσουμε και να την αιτιολογήσουμε λίγο περαιτέρω. Τέλος, και εδώ θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την εξέταση της ε, έκθεσης ΛΕΠΑΣ δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα διότι καθυστέρησε και η μετάφραση στα αγγλικά αλλά θα ήθελα να πω ότι πραγματικά ε, είναι πολύ καλή η ιδέα της ε, για ρήτρες grandfathering και θα ήθελα να τις εξετάσω. δεν είμαι βέβαια απόλυτα βέβαιη που μπορεί να μας οδηγήσουν. Ευχαριστώ κύριο Σιμάνσκι για τέσσερα λεπτά. Είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό πολύ πρόσφατα. Μιλήσαμε για την σταθερότητα από πολιτικής απόψεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την αξιοπιστία και βεβαίως τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία αυτών των αποφάσεων. Από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα, η εντύπωση που έχουμε είναι ότι οπισθοχωρούμε. Δηλαδή επιστρέφουμε στο παρελθόν και ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόμαστε το θέμα αυτό ίσως θα έπρεπε να αλλάξει. Στην Πολωνία οι επιχειρηματίες έχουν κάνει πολύ σοβαρές επενδύσεις Και αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα είναι ότι υπάρχει πιο απλοποιημένη διαδικασία με λιγότερη γραφειοκρατία. Εμείς σαφώς και μπορούμε να πούμε πολλά κατά αυτής της πρότασης, αυτής της πρωτοβουλίας, γιατί θεωρούμε ότι κατά κάποιο τρόπο έχουμε κάνει ήδη κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα ακυρώσουμε. Είναι σαφές από τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα ότι θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης της χώρας μου. Θα πρέπει σαφώς να δούμε το θέμα της έμεσης ε, αλλαγής της ε, χρήσης των εδαφών, της χρήσης της γης και την ίδια ώρα, καθότι ο στόχος μας είναι η μείωση των ε, αέριων του θερμοπικίου, ξέρουμε ότι σε πολλές χώρες η παραγωγή κάποιων ε, συγκεκριμένων φυτών σήμερα αφιερώνεται αποκλειστικά και μόνο στην παραγωγή βιοκαυσίμων και δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένες χώρες όπως τη Μαλαισία ή άλλες χώρες, αλλά οι αποφάσεις κάποιων ε, κρατών που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σίγουρα μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις και σε εμά. Επίσης σας μην ξεχνάμε και το θέμα της ε, μείωσης των ε, δασικών επιφανειών. Ξέρετε ότι μία τρίτη χώρα, μία χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να πάρει αποφάσεις που να επηρεάσουν και την δική μας εξάρτηση από αυτού του είδους τα καύσιμα. Υπάρχουν διάφορες παραγωγές που χρησιμοποιούνται σήμερα για την διάφορες καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παραγωγή βιοκαυσίμων όπως τα ζαχαρότεφλα. Ξέρουμε ότι η μείωση στην κατανάλωση ζάχαρης, παραδείγματο χάρη, είναι κάτι που οδήγησε προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά οι πολιτικές μας αποφάσεις, οι οποίες μας οδηγούν σήμερα στην εξέταση πιο προηγμένων βιοκαυσίμων, μιλάμε για δεύτερη και τρίτη γενιά βιοκαυσίμων, θα πρέπει να λάβει υπόψη της και τις τεχνικές ε, δυνατότητες αλλά και την ε, ανθρώπινη δραστηριότητα καθώς και τις επενδύσεις. Σήμερα υπάρχουν συγκεκριμένοι επιχειρηματίες που έχουν επενδύσει τα χρήματά τους σε κάποιο τομέα και κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς απολύτως καμία απόδοση. Ευχαριστώ πολύ. Ο η κυρία Κόπερτ, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγήτρια, την Κορίν Λεπάζ. Είναι πολύ ισορροπημένη η πρότασή της και νομίζω ότι είναι και μια πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση και επεξεργασία. Στηρίζω λοιπόν πλήρως τις προτάσεις της. Θεωρώ ότι και για τις μεταφορές θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πολύ σοβαρά και αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια και να μπορέσουμε να εξαλείψουμε συγκεκριμένες ε, γεωργικές πρώτες ύλες, γιατί σήμερα βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ σοβαρή ε, σε ένα πάρα πολύ σοβαρό ανταγωνισμό θα έλεγα μεταξύ των καλλιεργειών για την παραγωγή ειδών διατροφής και αυτών που προορίζονται για τα βιοκαύσιμα. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να στηρίξουμε και να επιλέξουμε βιώσιμα μοντέλα και να αναρωτηθούμε αν τα επιστημονικά αποτελέσματα που διαθέτουμε είναι επαρκή. Είναι αρκετά σοβαρά και βάσιμα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να πάρουμε πολιτικές αποφάσεις βάσει επιστημονικών δεδομένων που δεν είναι επαληθευμένα και σίγουρα. Σας ευχαριστώ. Τα επόμενα ονόματα που έχω είναι Αγιούζο, Ιβκοσέ και έχω ξεχάσει και κάποιος άλλος, αλλά έχετε όλοι δύο λεπτά. Κύριε Γιούζο, ευχαριστώ πολύ. Θα εκμεταλλευτώ το χρόνο μου και θα κάνω μια-δυο γενικές παρατηρήσεις ε, αφού ευχαριστήσω την ησυχήτρια και τους κοιόδες εισηγητές. Καταρχά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 10 χρόνια, εγώ ήμουν εισηγήτρια για την πρώτη οδηγία για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια ε, ω μέλο επιτροπή βιομηχανία. Ε, το Κοινοβούλιο ήταν υπέρ των βιοκαυσίμων, διότι τα βιοκαύσιμα αποτελούσαν καλή λύση για την γεωργική παραγωγή, διότι ήταν πολύ καλά, ε, ε, καλή δυνατότητα για τη διαφοροποίηση τη παραγωγή ενέργεια και φυσικά διότι έπρεπε να υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας. το 2008 έγιναν δεσμευτικοί οι στόχοι και έκτοτε έγιναν πάρα πολλές επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τους κανόνες ε, τους οποίους καθορίσαμε τότε. Υπάρχουν πάρα πολλές επενδύσεις και πάρα πολλές θέσεις εργασίας τις οποίες δεν μπορούμε πλέον ούτε να τις αμφισβητήσουμε αλλά ούτε και να τις θέσουμε κινδύνο. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε και να αποδείξουμε ότι όντως κάναμε καλή πολιτική. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου και δεν θα πρέπει να βασανίσουμε, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τον όρο, τις επιχειρήσεις που επέλεξαν να επενδύσουν σε βιοκαύσιμα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να θέλουμε να ξεχάσουμε μία νυχτή του στόχους που έχουμε για τα βιοκαύσιμα πρώτης γενεάς ε, και για βιοκαύσιμα τα οποία αποκαλούμε τώρα συμβατικά χωρίς ε, ε, να τους δώσουμε μια δυνατότητα. Θα πρέπει να κάνουμε επενδύσεις σε προηγμένα βιοκάσιμα δεύτερης και τρίτης γενεάς, αλλά θα πρέπει να κερδίσουμε και από τις επενδύσεις που έγιναν στα πρώτης γενεάς. Τώρα, για τους συντελεστές ILEC, ε, τα μοντέλα αυτά δεν έχουν επιστημονική βάση. Πρόκειται για ένα επιπλέον διοικητικό άχθος το οποίο δεν μπορεί να βοηθήσει ε, την παραγωγή βιοκοψίμων και είναι κάτι το οποίο ναι, μεν πρέπει να συνεχίσουμε να μελετούμε, αλλά δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε. Δύο λεπτά μόνο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είναι εντυπωσιακό το ότι εδώ αυτή η έμεση αλλαγή της χρηστικής, αυτός ο συντελευτής, ε, ήδη αμφισβητείται από αυτούς που αρχικά τον πρότειναν. Πρέπει λοιπόν πραγματικά να δούμε το κατά πόσο υπάρχει αξιοπιστία πριν προχωρήσουμε στη δεύτερη και τρίτη γενιά και πριν προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε επενδυτές για αυτές τις μελλοντικές παραγωγές. Θα πρέπει επίσης να δούμε αν θα συνεχίσει να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς άλλους τομείς και προς την παραγωγή ε, ειδών διατροφής αλλά και προς άλλους τομείς όπως η χημεία παραδείγματος χάρη. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να δούμε τις επιπτώσεις για άλλες γειτονικές περιοχές. Επίσης όσον αφορά την εκμετάλλευση και τη χρήση της γης. Πώς επηρεάζει δηλαδή αυτή η νέα παραγωγή την γεωργική παραγωγή, την εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής και έχω την εντύπωση ότι ο τομέας της ενέργειας είναι πολύ περιορισμένος, δεν μπορούμε δηλαδή όλα να τα θυσιάσουμε. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να δούμε τον ε, παράγοντα της βιοποικιλομορφίας. Θα πρέπει αυτή η παραγωγή να προσθέτει κάτι, όχι μόνο να καταστρέφει υπάρχουχες καλλιέργειες. Και βεβαίως ένας άλλος τομέας με τον οποίο μπορεί να είναι πολύ ε, ανταγωνιστική αυτή η παραγωγή είναι οι ζωοτροφές αλλά και άλλες μορφές παραδοσιακής ε, γεωργικής παραγωγής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζέμπερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ πρόκειται για την αξιολόγηση κάποιων ε, νομοθετικών κειμένων μιας νομοθεσίας του 2008. Καλούμαστε να δούμε τα αποτελέσματα αυτών των αποφάσεων βλέπουμε ότι μιλάμε για μια τεράστια εδαφική έκταση που κάθε χρόνο βγαίνει από την αγροτική καλλιέργεια και παραγωγή πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια εκτάρια το χρόνο και αυτό είναι εντυπωσιακό. Αυτό που επίσης θα πρέπει να αξιολογήσουμε είναι αν αυτές οι εκτάσεις χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά είχαμε προβλέψει. Ξέρετε παραδείγματος χάρη και στο παρελθόν είχε γίνει τέτοια μεταστροφή παραγωγής, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα ε, εγκατάλειψη εγκαταστάσεων, υποδομών, οικονομική ύφεση στις περιοχές καθότι οι επόμενες επενδύσεις δεν προσελκύονται άμεσα. Επίσης έχουμε και ε, περιβαλλοντολογικές αλλά και κλιματικές επιπτώσεις. Δεν δικαιολογείται δηλαδή εδώ αυτή η παραγωγή εάν δεν τη δούμε πολύ πιο ολοκληρωμένα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε, παραδείγματο χάρη, την βιωσιμότητα αυτών των επενδύσεων και θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους ε, από νομικής απόψεως για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία όντως αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Είναι αμφισβητούμενα πολλά από τα σημεία αυτής της πρότασης. Επιτρέψτε μου τελειώνοντας να πω ότι υπάρχουν και κάποια οικονομικά αν θέλετε προβλήματα και αδυναμίες. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτή η έμεση αλλαγή της χρήσης γης συμπεριλαμβάνει αρκετές μελέτες όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις που δεν συμπεριλαμβάνει αυτή η πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής για δύο λεπτά, κύριο Στέμπερ. Ευχαριστώ. Εμείς ε, αποφασίσαμε πριν από δύο εβδομάδες ε, στην Επιτροπή μας και ήμασταν πάρα πολύ, αν θέλετε, ευκριτικοί στην πρότασή μας. Δεν καταλάβαμε ακριβώς ε, τι έγινε με την πρώτη γενιά βιοκαυσίμων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε τότε εκφράσει την επιφύλαξή του. Είχαμε πει πρέπει να είμαστε προσεκτική. Είχαμε θέσει σαν στόχο το 10% όχι για τα βιοκαύσιμα αλλά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γενικότερα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχουν προβλήματα και κάποιες συγκρούσεις και ανταγωνιστικές, ε, αν θέλετε, προσεγγίσεις. Τα βιοκαύσιμα, ναι, κάλυψαν κάποιες ε, ελλείψεις. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι υπάρχουν σήμερα εκτάσεις που δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι χρησιμοποιούνται με τον πιο ε, χρήσιμο από οικονομικής απόψεως, από κοινωνικής απόψεως τρόπο. Ευχαριστώ πολύ ε, τους ε, εισηγητές από την Επιτροπή Ήτρε, παραδείγματος χάρη με τον οποίο συνεργαστήκαμε πολύ θετικά. Θα πρέπει να εντοπίσουμε όμως καλύτερα πού υπάρχουν αδυναμίες. Παραδείγματο χάρη, ο κατάλογος των πρώτων υλών που συμπεριλαμβάνει εδώ η πρόταση. Και θα σα δώσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Όπως έχει σήμερα η πρόταση και ο κανόνας, οδηγούμαστε σε ένα αδιέξοδο. Δηλαδή, βλέπετε ότι τα φυτικά έλαια, παραδείγματο χάρη, φοινικέλαιο έλαιο και άλλα, θα μας οδηγήσουν σε περισσότερες εισαγωγές ζωοτροφών από την Αμερική. Καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι ένα πάρα πολύ ε, αρνητικό αποτέλεσμα μιας ε, αρχικά θετικής ιδέας, κάτι που θα μας οδηγήσει σε χρησιμοποίηση για ε, διαφορετικούς σκοπούς αυτών των πρωτεϊνών παραδείγματο χάρη, πρωτεϊνών που σίγουρα είναι πολύ χρήσιμες, οι οποίες όμως σήμερα θα χρησιμοποιηθούν για βιοκαύσιμα, κάτι το οποίο ανατρέπει τελείως την παραδοσιακή τους χρήση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Να σας ευχαριστήσω επίσης και για όλα τα σχόλια τα οποία ακούσαμε σήμερα. Σίγουρα το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο από οικονομικής, τεχνολογικής, περιβαλλοντικής πλευράς. Νομίζω ότι ε, η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνεται σε τρία πράγματα. Να μειωθούν οι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου, να έχουμε μια βεβαιότητα όσον αφορά τι επενδύσει και να καταφέρουμε να διαχειριστούμε ένα σωστό σύστημα καταγραφή. Αυτό το κάναμε με το 5%, με το νότατο όριο του 5% και το πετύχαμε επίσης και με την ενθάρρυνση των μελλοντικών επενδύσεων σε νέες μορφές ενέργειας. Και χρησιμοποιούμε επίσης και διάφορους παράγοντες προκειμένου να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις έμεσες επιπτώσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να δούμε άμεσα. Δεν θα συμφωνούσαμε όσου λένε ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα επιστημονικά δεδομένα, ότι δεν είναι βάσιμα αυτή τη στιγμή. Εμεί σαφώ έχουμε χρησιμοποιήσει κάποια μοντέλα. Θεωρούμε πάντω ότι ε, τα μοντέλα αυτά έχουν μια σωστή επιστημονική βάση, έχουν επαληθευθεί πολλές φορές και μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά. Επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση έχουμε και την αρχή της προφύλαξης. Επομένω, ακόμα και αν υπάρχει ακόμα και ένας κίνδυνος μπορούμε να λειτουργήσουμε βάσει της αρχής της ε, πρόληψης που χρησιμοποιείται στα πλαίσια του μοντέλου. Όσον αφορά τώρα τις διάφορες ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί για την έκθεση αυτή. Σαφώς είμαι υπέρ οποιασδήποτε βελτίωση των ορισμών, οτιδήποτε μπορεί να βελτιώσει τους ορισμούς και μπορεί να βελτιώσει τελικά την ποιότητα της πρότασης είναι καλοδεχούμενο. Θεωρούμε επίσης ότι θα πρέπει να επεκταθεί το όριο του 6% μετά το 2020, αν μπορούν τελικά οι φορείς να ανταποκριθούν στο σύστημα το οποίο προβλέπεται στην έκθεση όσον αφορά τα κριτήρια βιωσιμότητα. Νομίζω ότι αν έχουμε καλύτερου ορισμού θα καταφέρουμε να έχουμε και καλύτερα τέτοια κριτήρια. Όσον αφορά τώρα τη συμπερίληψη του στελεστή Άιλουκ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε σωστή καταγραφή τη έμεση αλλαγή τη χρήση γη και αν γίνουν σωστέ μετρήσει θα καταφέρουμε να πάρουμε και σωστά αποφάσει. Ο παράγοντα αυτό πάλι βασίζεται σε σωστά επιστημονικά δεδομένα. Όπω βλέπετε όμω και από την έκθεση αντικτύπου, θεωρούμε ότι θα πρέπει στην τελική πρόταση να ε, συμπεριληφθούν παράγοντες στα κριτήρια βιωσιμότητος, γιατί θεωρούμε ότι αυτό θα έχει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις στην ε, βιομηχανία και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι σε μια πρώτη φάση δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όσον αφορά το grandfathering της ρήτρες κεκτημένων δικαιωμάτων, και αυτές αναφέρουμε στην πρότασή μας. Βλέπουμε επίσης ότι ε, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ανώτατα όρια εμείς θεωρούσαμε ότι τα όρια αυτά θα έπρεπε να υφίστανται, αλλά νομίζουμε ότι τουλάχιστον στην πρόταση γίνονται κάποιες, έχουν υποβληθεί κάποιες τροπολογίες για να απομακρυνθούν. Στα παραρτήματα έχουμε και μία σειρά από φυτίες και τρόφιμα για τα οποία υπάρχει πολλαπλή προσμέτρηση. Είναι μια εργασία που ήδη έχουν ξεκινήσει τα κράτη-μέλη. Θεωρούμε ότι ε, η λίστα αυτή τη στιγμή, ο κατάλογο είναι πλήρη διεξοδικό. απαιτήθηκε πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να καταρτιστεί. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο με την προσμέτρηση τη διπλή ως την τετραπλή να καταφέρουμε να προωθήσουμε καλύτερα την ανάπτυξη των νέων αυτών βιοκαυσίμων. Θέλουμε να συνεργαστούμε περισσότερο με την εισηγήτρια και του σκιώδη εισηγητέ για να βελτιώσουμε όλε τι πτυχέ τη πρόταση και συνεργαζόμαστε επίση και με τι υπόλοιπε έξι επιτροπέ οι οποίε γνωμοδοτούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά δεν ήταν ο Χάνης Φωνστέιν. Το καταλάβατε. Έχω τρεις συναδέλφους. Χίμπνερ, Μπάνκι και Κωσέ, οι οποίοι έχουν ζητήσει το λόγο. Και κατόπιν εισηγήτια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, πραγματικά ήθελα να λάβω το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προτείνει αυτόν τον νέο συντελεστή iLook. Αλλά εδώ και το ερώτημα κατά πόσον η παραγωγή βιοκαυσίμων αποτελεί απειλή για την βιοπικιλότητα. Ίσως με την παραγωγή βιοκαυσίμων να στερούμε τα δάση από το περιβάλλον ή από γεωργικές εκτάσεις στις οποίες παράγονται τρόφιμα. Ισχύει όμως αυτό. Εγώ δεν νομίζω διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερεπάρκεια τροφίμων ε, στις γεωργικές περιοχές και το πρόβλημα είναι αν θα μπορέσουμε να τα εξάγουμε εκτός Ευρώπης. Και θα ήθελα να σκεφτούμε και το εξής. δεν υπάρχει σταθερότητα ως προς το δίκαιο. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι θα υπάρχει μακροπρόθεσμη σαφήνεια, διότι τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται για ένα-δυο χρόνια, ε, δεν γίνεται κατάλληλος προγραμματισμός και δεν γίνεται ε, προγραμματισμός μόνο πενταετίας, ε, γίνεται προγραμματισμός μακροπρόθεσμος. Και το ίδιο ισχύει και για τα μακροπρόθεσμα προγράμματα επενδύσεων για τους γεωργούς. Θα πρέπει λοιπόν εμείς ως νομοθέτες να αναπτύξουμε τον τομέα των βιοκαυσίμων στην Ευρώπη και αυτό φυσικά να μας οδηγήσει σε διαφοροποίηση της χρήσης διαφόρων ενεργειακών πηγών, να μπορέσουμε να έχουμε κατάλληλα προϊόντα για τη γεωργία και επίσης να να έχουμε και μία εναλλακτική λύση για την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών. Δεν γίνεται να τα πετάξουμε όλα στα σκουπίδια και θα ήθελα να γνωρίζω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που γνωρίζει πως έχει κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και οι γεωργοί μας πίστευσαν, οι επενδυτές μας πίστεψαν. Πραγματικά όλα αυτά θα τα πετάξουμε ε, στα σκουπίδια και θα τους πούμε ότι όλα όσα κάνατε δεν αξίζει τίποτα γιατί αύριο θα αρχίσουμε να ε, φυτεύουμε καρότα και σμέουρα εδώ στους ε, γεωργικές εκτάσεις. Πρέπει να είμαστε σαφείς αυτά που κάνουμε γιατί αλλιώ θα γίνουμε περίγελος. Ευχαριστώ πολύ κύριο Μπάνκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με αυτά που είπε μόλις τώρα η κυρία Χιούμπνερ, θα ήθελα να πω ότι αν κοιτάξει κανείς τις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, την Ουγγαρία, είμαστε λίγο καθυστερημένοι σε σχέση με την καλλιέργεια για την παραγωγή βιοκαυσίμων δεύτερης και τρίτης γενιάς. Και αν κοιτάξετε πολύ συγκεκριμένα την Ουγγαρία, θα σας πω ότι κατά μέσο όρο παράγουμε 3 ή 4 εκατομμύρια τόνους δημητριακών σε σχέση με αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για την χώρια <clears throat> παραγωγή μας. Έχουμε εξάλλου μεγάλη δυσκολία στο να εξάγουμε αυτή την παραγωγή και να αποθηκεύσουμε αυτά τα προϊόντα. Αυτό μας ε, οδηγεί στην χρησιμοποίηση αυτής της παραγωγής ε, για βιοκαύσιμα. Και αυτό είναι κάτι που αποτελεί για μας μια εξαιρετική λύση. Έχουμε τρεις μονάδες οι οποίες επιτρέπουν στους ε, καλλιεργητές, στους γεωργούς να προμηθεύουν αυτήν την παραγωγή. Εάν όμως τελικά αλλάξουν τα ποσοστά, για μας ε, κινδυνεύουν όλοι αυτοί οι παραγωγοί να βρεθούν σε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Μόλις ξεκινήσαμε την παραγωγή βιοεθανόλης στη χώρα μας, κάτι που πραγματικά έχει αποδειχθεί πάρα πολύ καλή ευκαιρία για την διοχέτευση αυτής της παραγωγής. Ο κύριος Κωσέ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρω την κυρία Λεπάζ για την πολύ πλούσια έκθεσή της. Θα ήθελα να πω όμως ότι πρέπει να είμαστε αντίθετοι με τα βιοκαύσιμα και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Πρέπει να σταματήσουμε την παραγωγή του. Αυτό που ακούω όμως μου φαίνεται παράλογο. Ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια. Ναι, σήμερα διαπιστώνουμε και περιβαλλοντολογικά και άλλου είδου προβλήματα, στον τομέα τη υγεία παραδείγματο χάρη. Παρ' όλα αυτά όμω, θα μειώσουμε την παραγωγή, θα συνεχίσουμε όμω, Όχι. Πρέπει πραγματικά να σταματήσουμε το συντομότερο δυνατόν, όχι μόνο για θέματα υγείας, όχι μόνο για θέματα περιβάλλοντος, αλλά και για θέματα ενέργειας και για οικονομικές αιτίες. Αν κοιτάξουμε πραγματικά τα επιστημονικά δεδομένα, θα δούμε ότι δεν είναι θετικό το αποτέλεσμα, το ενεργειακό αποτέλεσμα της ε, παραγωγής βιοκαυσίμων. Και η βιοεθανόλη και τα άλλα βιοκαύσιμα σαφώς έχουν αρνητικό αποτέλεσμα ενεργειακό. Καταναλώνουν δηλαδή περισσότερη ενέργεια για την παραγωγή τους από ό,τι τελικά παράγουν. Τα βιοκαύσιμα δεν πρόκειται λοιπόν ποτέ να είναι αποτελεσματικά. Και αυτό που μας λένε τώρα είναι ότι ίσως η δεύτερη γενιά βιοκαυσίμων να είναι αποτελεσματικά. Αυτή δηλαδή η γενιά στην οποία χρησιμοποιούμε τους καρπούς, τους σπόρους αυτών των φυτών. Είναι παράλογο. Είδαμε ότι το αποτέλεσμα πάλι δεν είναι θετικό. Ευχαριστώ πολύ. μπορείτε να πάρετε το λόγο. Έχουμε μικρόφωνα, μεγάφωνα, ηχεία. Θα δώσω το λόγο στην ηθηγητρία. Κυρία Λεπάζ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο. Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή και θα ήθελα να σας πω πολύ απλά ότι μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε για να αποφύγουμε την ουσία. Σκοπός μας είναι η μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου και μπορεί να μην θέλουμε να το διαπιστώσουμε, αλλά τελικά κάτι τέτοιο δεν το επιτυγχάνουμε. Όλοι όσοι θα συνεχίσουν σε αυτόν τον τομέα και όλους όσους θέλουν να τηρήσουμε αυτό το στόχο, θα πρέπει τουλάχιστον να τους πούμε την αλήθεια. Τώρα, όσον αφορά αυτό το συντελεστή για την ε, έμεση αλλαγή χρήση της επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι δεν είναι ευρωπαϊκό μοντέλο. Εφαρμόζεται ήδη στην Καλιφόρνια, στις Ηνωμένε Πολιτείε. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι η επιστήμη δεν είναι αξιόπιστη, δεν είναι αρκετά σίγουρη Παρ' όλα αυτά κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε μία απόφαση για να μην παραμείνουμε στο σημερινό σύστημα. Κάτι που δεν θα ήταν σωστό κατά την άποψή μου. Δεν μπορούμε δηλαδή επάπειρο να επικαλεστούμε αυτήν την επιστημονική έλλειψη σιγουριάς για να μην κάνουμε τίποτα. Τρίτον, δεν μπορώ να σας αφήσω να επαναλαμβάνετε ότι η πρότασή μου θα οδηγήσει στο κλείσιμο επιχειρήσεων και στην απώλεια θέσεων απασχόλησης. Αυτό δεν ισχύει καθότι υπάρχει ένα σύστημα που θα συνεχίσει να ισχύει με μεγάλη γενεοδορία για τους ε, γεωργούς, για τους παραγωγούς βιοκαυσίμων. Επαναλαμβάνω ότι αυτό κοστίζει 10 δις κάθε χρόνο και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ με έναν τρόπο πολύ πιο αποτελεσματικό. Παρ' όλα αυτά δεν το προτείνω. Προτείνω να διατηρηθούν οι επενδύσεις Θα πρέπει παρόλα αυτά να γνωρίζουμε αυτά τα στοιχεία, αυτούς τους αριθμούς. Άκουσα επίσης πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε όσον αφορά τον ε, αγροτικό στόχο. Δεν πρόκειται όμως για γεωργική νομοθεσία. Πρόκειται για μια νομοθεσία που έχει σαν στόχο την ποιότητα των καυσίμων και την μείωση των ε, αερίων θερμοκηπίου. Βεβαίως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τα συμφέροντα των αγροτών. Αυτή όμως η νομοθεσία δεν έχει αυτό το αντικείμενο. Αν μου πείτε ότι ο σκοπός αυτής της νομοθεσίας είναι να επιδοτήσουμε τη γεωργία και όχι να προστατεύσουμε το περιβάλλον, τότε ας είμαστε ειλικρινείς και ας μην κρυβόμαστε πίσω από άλλους στόχους που είναι η αλλαγή του κλίματος, παραδείγματο χάρη. Σας προτείνω λοιπόν κάτι που μου φαίνεται ισορροπημένο, γιατί θεωρώ ότι λαμβάνουμε υπόψη μας τα συμφέροντα αυτών που έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις, τα συμφέροντα των γεωργών, αυτών που παράγουν βιοκαύσιμα. Κοιτούμε όμως και αυτήν την παραγωγή η οποία δεν είναι βιώσιμη. Εγώ δεν πήγα στη Μαλαισία, αλλά Πρέπει να σας πω ότι συνάντησα εκπροσώπους των Ιθαγενών πληθυσμών στη Μαλαισία, οι οποίοι μου περιέγραψαν την συμπεριφορά και τις πρακτικές των επιχειρήσεων, οι οποίοι καίνε την γη, περιορίζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των ε, μικροκαλλιεργητών και κατόπιν καταστρέφουν τις καλλιέργειες με σκοπό να παράγουν φινικέλαιο και άλλες καλλιέργειες που έχουν σαν αποκλειστικό σκοπό τα βιοκαύσιμα. Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζουμε βεβαίως την ε, συζήτηση. Το θέμα είναι ανοιχτό. Περιμένω όλες τις προτάσεις των σκιωδών εισηγητών. Ο κύριος ε, Βλευκάντρας σαφώς και είναι διατεθειμένος για περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων και εγώ το ίδιο και ελπίζω να φτάσουμε σε μια ισορροπημένη πρόταση η οποία θα λαμβάνει υπόψη της όλες αυτές τις προτεραιότητες. Ευχαριστώ πολύ. Κορίν Λεπάς. 27 Μαΐου είναι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. και θα συζητήσουμε εδώ στις 19 και 20 Ιουνίου έτσι ώστε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Σεπτέμβριο. Ψηφίζουμε στην Επιτροπή τον Ιούλιο. Προωρούμε τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της της διάταξης που είναι το σημείο 6. Η συγητής, ο κ. Μπαρτολότσι, καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη βιοκαινοτομία για την Ευρώπη. Ο Όποιος θέλει να εγκαταλείψει την αίθουσα παρακαλώ πολύ να το κάνει με ησυχία. Und Ίσως οι συζητήσεις ε, για το ILOC μπορούν να συνεχιστούν εκτός της ε, αίθουσας. Θέλουμε να ακούσουμε τον εισηγητή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους όσους ε, συνεισέφεραν στο θέμα αυτό για τη βιοοικονομία. Σήμερα, πέρα από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, θα ήθελα εντάχει να σας περιγράψω τη θέση μου σε γενικές γραμμές και το τι σκοπεύω να λάβω υπόψη ε, όταν θα εξετάσουμε το ζήτημα. Όπως θα γνωρίζετε, κατατέθησαν μια σειρά από τροπολογίες, ε, αρκετές τροπολογίες ε, τολμώ να πω, 100 τροπολογίες και επομένως έπρεπε να καταλήξουμε σε κάποιους συμβιβασμούς. Όσον αφορά τις γενικές γραμμές τις οποίες θα ήθελα να ακολουθήσω, ε, θα μπορούσα να δεχτώ όλες τις τροπολογίες οι οποίες ε, κάνουν κάποιες τροποποίησεις ή προσθήκες οι οποίες ε, προσφέρουν περισσότερη σαφήνεια στο αρχικό κείμενο και ενισχύουν με θετικό τρόπο κάποιες έννοιες οι οποίες έχουν ήδη εκφραστεί ή εισαγάγοντας κάποιες καινούργιες σεβόμενοι πάντα την γενική τοποθέτηση ε, της Συμφωνία με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα δεχτώ δηλαδή τροπολογίες ε, οι οποίες επισημαίνουν τη σημασία της περιφερειακής διάσταση και στόχο έχουν να ε, εδρεώσουν την ε, βελτίωση του γεωργικού και βιομηχανικού τομέα λαμβάνοντας υπόψη του ταυτόχρονα και την βιοπικιλότητα. Όσον αφορά το έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. συμφωνώ με αυτέ που ζητούν να υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για την υποστήριξη τη βιοοικονομία από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την εισαγωγή μέσων τα οποία ολοκληρώνουν το πρόγραμμα δράση ε, που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω για παράδειγμα την ενιαία θηρίδα πληροφοριών για πρωτοβουλίε, οι οποίε συνδέονται με τη βιοοικονομία. Όσον αφορά την ενίσχυση των αγορών ε, και τη δέσμευση των διαφόρων μερών, συμφωνώ με τι τροπολογίε, οι οποίε επιβεβαιώνουν πόσο πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότηση τη βιοοικονομία στα πλαίσια προγραμμάτων και ε, κοινοτικών πολιτικών και ε, να υπάρχουν ευρωπαϊκές διαδικασίες ε, έγκριση συγκεκριμένων ε, προϊόντων που επιβεβαιώνουν πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αγορά. Και θα πρέπει να υπάρχει φυσικά και βιώσιμη ανάπτυξη της βιομάζας. Δεν συμφωνώ όμως με τροπολογίες που εμένουν μόνο στις αρνητικές πτυχές της βιοοικονομίας χωρίς ε, να κάνουν καμία επικοδομητική πρόταση ή που ε, κάνουν κάποιες υποδείξεις οι οποίες είναι περιτές και επαναλαμβάνουν κάποιες έννοιες τις οποίες έχουμε πει επανειλημμένως σε άλλα σημεία του κειμένου. Ε, και υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ήδη υποθεί. Ε, όπως επίσης θεωρώ ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω τροσοπολογίε, οι οποίες υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογή ε, του θέματος που εξετάζουμε, ούτε και τροποποιήσεις οι οποίες στόχο έχουν να διαγράψουν κάποια στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι είναι θεμελιώδη σημασία. Αναφέρομαι για παράδειγμα στον ε, πίνακα για τις ε, βιομηχανίες και κάποιες βιομηχανικές δραστηριότητες οι οποίες δεν θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να έχουμε επενδύσεις σε βιομηχανικές εμπορική κλίμακα, ε, σε εμπορική κλίμακα συγγνώμη, για τη βιοοικονομία και επίσης την άρση κάποιων γραφειοκρατικών οχλήσεων για την ανάπτυξη συγκεκριμένων μέτρων βιοοικονομίας, όπως επίσης και τα απαραίτητα φορολογικά μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα για να υπάρχει κατάλληλη έρευνα στον τομέα και να υποστηρίξουν όλους όσους εφαρμόζουν στην πράξη αυτά τα κατάλληλα αποτελέσματα, δηλαδή τη βοήθεια προς επιχειρώσει. επιχειρώσεις, ε, ε και να υπάρχουν και κατάλληλες ε, δυνατότητες στην αγορά για τη βιομάζα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ε, είμαι διατεθειμένος βέβαια να ακούσω όλες τις απόψεις και να απαντήσω και σε πιθανές ερωτήσεις ε, που αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα. Ευχαριστώ. Eh. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Μέρκης, και να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μπαρτολότσι γιατί ξεκαθάρισε την άποψή του. Έχουμε εξετάσει ήδη την πρόταση αυτή στα πλαίσια της Επιτροπής. Έχουμε μιλήσει εκτενώς για τα ζητήματα της βιοοικονομίας. Έχουμε δει ότι τα πλονεκτήματα είναι πάρα πολλά. Έχουμε δει ότι τα συμφέροντα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και πιστεύω ότι η βιοοικονομία έχει λαμπρό μέλλον μπροστά της. Μπορεί να αποτελέσει πηγή ενέργειας, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα καινοτόμα προϊόντα σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Τώρα, από πλευράς αρνητικής, αρνητικού αντικτύπου, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες. Θεωρώ ότι πολλές φορές προσεγγίζουμε την βιοοικονομία ως το μοναδικό μέσο το οποίο έχουμε μπροστά μας. Ουσιαστικά μπορεί εντελώς να υποκαταστήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πορεύουν από τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία όπως γνωρίζετε σπανίζουν όλο και περισσότερο. Θα πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι η βιοοικονομία πρέπει να συνδέεται και με μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς επίσης και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί ουσιαστικά να υπάρξει στο μέλλον. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε ένα είδος ιεραρχίας, αυτή την διαδοχική λεγόμενη χρήση της βιομάζας. θα πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη βιομάζα καταρχάς μόνο εκεί που έχει την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Γιατί φοβάμαι ότι καταναλώνεται αυτή τη στιγμή σε ένα μεγάλο ποσοστό βιομάζας. Αντί να χρησιμοποιείται με τρόπο αποτελεσματικό. Πιστεύω λοιπόν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βιομάζα σε συνδυασμό με άλλες πηγές ενέργειας, χωρίς να αντικαθιστούμε τις κλασικές πηγές ενέργειας με τη βιομάζα. Ελπίζω ότι ο συγητής στα σημεία αυτά τα οποία έχω θέσει θα με υποστηρίξει. Επίσης πρέπει να διασυνδέσουμε, όπως σας είπα, τη βιοοικονομία με άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα η αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων και το καθεξής. Και επίσης θα πρέπει να συνδεθεί περισσότερο με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, καθώς επίσης και με το 7ο πρόγραμμα έρευνας. Νομίζω ότι όλοι μας συμφωνούμε ότι η ενθάρρυνση περισσότερο της έρευνας στον τομέα αυτό, είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω όμως παράλληλα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που απορρέουν από τη βιομάζα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποφύγουμε μελλοντικά προβλήματα εφαρμογής της βιομάζας στην πράξη, στην οικονομία δηλαδή. Μία τελευταία παρατήρηση καλύτερη χρήση της γης και των υδάτων, καλύτερο συντονισμό ως προς τη χρήση αυτή, καθώς επίσης και μία πιο έντονη κοινωνική εταιρική ευθύνη, που νομίζω ότι και στον τομέα αυτό της βιομάζας και της βιοοικονομίας ισχύει, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο εξ ονόματος του συνάδελφου Τζαμπάνη, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί για τη σημερινή συζήτηση και ζητά συγγνώμη ε, για την απουσία του. Θα πω εγώ δύο λόγια εκ μέρους του. Με την ε, γνωμοδότηση προσπαθεί ο κύριος Μπαρτολόξη να ε, ενισχύσει την ε, ανακοίνωση για την καινοτομία για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι πρέπει να αναζητήσουμε νέους τρόπους ε, βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, επομένως θα πρέπει να λάβουμε μέτρα για να επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες και να δημιουργήσουμε και δυνατότητες που θα έχουν μακροπρόθεσμα ωφέλη για την οικονομία. Όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, υπάρχουν πολλές τροπολογίες που αναφέρουν ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διάρκεια και θεωρούμε ότι το κριτήριο της διάρκειας θα πρέπει να είναι πολύ σημαντικό για την ε, βιομάζα και για την ε, τρέχουσα πολιτική της κατασπατάλησης των πόρων μας. Θα πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και να ε, προσπαθούμε να έχουμε και βασική έρευνα για τα θέματα αυτά. Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις για να βελτιώσουμε το ρόλο των ηγετικό που έχει η βιομηχανία και θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τη δυνατότητα των μεταφορών, την κατάλληλη ε, δυνατότητες επιμελητίας και αποθήκευσης. Όσον αφορά τώρα για τις ε, τροπολογίες που αφορούν για τη χρήση της μειομάζας, εμείς ε, υποστηρίζουμε τη χρήση της ε, τεχνολογίας τη διαδοχική τεχνολογία και τη βιομάζας η οποία θα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς και θα πρέπει να μπορούμε να δούμε πώς μπορεί να βελτιώσει τα οικοσυστήματα. Όσον αφορά τώρα τις επιχορηγήσεις, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν επιδοτήσεις οι οποίες ενθαρρύνουν τη μη αποτελεσματική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε υποβάλει λοιπόν την ε, ε τροπολογία 97 η οποία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει αυτή την κατασπατάλωση. Υπήρχε αντίστοιχη αντίστοιχη τροπολογία στο 7ο πρόγραμμα ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άιχου τώρα έχει το λόγο, ο οποίος αντικαθιστά την κυρία του Χάση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Χάση δεν μπορεί να είναι σήμερα το απόγευμα εδώ πέρα και σας ζητά συγγνώμη. Μπορεί ότι βέβαια το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μπαρτολότση, εξ ονόματος κυρίας Χάση λοιπόν, για την έκθεση την οποία έχει εκπονήσει. Ορισμένες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω, οι οποίες συνάδουν με αυτά τα οποία είπαν οι υπόλοιποι συνάδελφοι, οι σοσιαλιστές για παράδειγμα. Νομίζω ότι όλο και περισσότεροι βλέπουμε ότι όντως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό στη βιοοικονομία, επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποια στρατηγική ακολουθούμε για την αντικατάσταση των ορεικτών καυσίμων από τη βιομάζα και ποιε είναι οι ενδυνάμει ε, πιθανότητες οι οποίες ε, εμφανίζονται στο μέλλον. Θα πρέπει να γίνει αυτό με τρόπο αποτελεσματικό, βιώσιμο και να χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά τη βιομάζα Καταρχά, στα σημεία εκεί πέρα, στα σημεία εκείνα που έχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και μόνο μετά στου τομεί εκείνου που έχουν ε, μικρότερη προστιθέμενη αξία. Αυτό εννοούμε όταν, όταν λέμε χρήση διαδοχική. Ξεκινάμε δηλαδή από τα υψηλότερα επίπεδα τη πυραμίδα και κατεβαίνουμε σιγά σιγά στα χαμηλότερα. Να χρησιμοποιηθεί καταρχάς η βιομάζα μόνο εκεί που εντοπίζεται μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η βιομάζα στα σημεία εκείνα, στους τομείς εκείνους με χαμηλότερη προστιθέμενη αξία και μόνο σε ίστατο πλέον στάδιο θα πρέπει η βιομάζα να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στις μονάδες δηλαδή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαδοχική λοιπόν αυτή χρήση αποτελεί μια πολύ σημαντική πτυχή της βιοοικονομίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι θα υλοποιηθεί αυτή η διαδοχική χρήση. Και ξέρετε ότι η πρώτη συζήτηση που κάναμε στα βιοκαύσιμα ακριβώς αυτό καταδεικνύει. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για τη χρησιμοποίηση της βιομάζας στις μεταφορές, πράγμα το οποίο δεν είναι η πιο αποτελεσματική χρήση. Α είμαστε λοιπόν αρκετά επικριτικοί και αρκετά προσεκτικοί, α συνειδητοποιήσουμε ότι σε αυτό το στάδιο η Ευρώπη δεν είναι ακόμα πάρα πολύ αποτελεσματική στη χρήση βιομάζας που κάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πράσινους να εξασφαλίσουν ότι όντως θα έχουμε μια αποτελεσματική χρήση της βιομάζας σε ένα σύστημα διαδοχικής χρήσης. Θέλουμε να το δούμε αυτό στο τελικό κείμενο του ψηφίσματος αυτού. Κάποιες άλλες παρατηρήσεις αν πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, εμπορική χρήση της ε, βιοοικονομίας Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κάτι είναι εμπορικά διαθέσιμο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να υπάρχει μια χρηματοδοτική υποστήριξη προς αυτό. Αν θέλουμε να υποστηρίξουμε τη βιομηχανία προκειμένου να αναπτύξει κάποια προϊόντα και υπηρεσίες σε προεμπορική φάση, τότε νέα υπάρχει χρηματοδοτική υποστήριξη, αλλά όχι χρηματοοικονομική υποστήριξη για την εμπορική φάση. Γιατί στην περίπτωση αυτή δεν θα μιλούσαμε για εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες. Όσον αφορά τι συμπράξει δημοσίου ιδιωτικού τομέα, ναι, μπορεί να υπάρχει πάλι μια υποστήριξη. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλε αυτέ οι εφαρμογέ τη βιομάζα θα πρέπει να γίνονται με τρόπο βιώσιμο. Διαφορετικά θα συναντήσουμε τα ίδια προβλήματα που έχουμε τώρα με τη χρησιμοποίηση βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών. Και αυτό το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε είναι η όλη, όλη συζήτηση για την βιοοικονομία να έχει τελικά την ίδια μοίρα με τα βιοκαύσιμα. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια τόσο αρνητική εικόνα για τη βιοοικονομία που κανείς τελικά δεν θα τη θέλει στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η προσέγγιση μας να είναι βιώσιμη σε κάθε περίπτωση. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά και το χένιο τη επιτυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι. Κατόπιν, ποιο έχει ζητήσει το λόγο, η Επιτροπή. Όχι, κανείς άλλος δεν ζητάει το λόγο. Η Επιτροπή λοιπόν. Έχετε το λόγο. Καλό σας απόγευμα. Και εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Στηρίζουμε την τροπολογία 40 που αναφέρεται στην βιοοικονομία και το παρατηρητήριο καθώς και την Επιτροπή για την βιοοικονομία. Πρόκειται για πολύ σημαντικά όργανα, φορείς όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για την βιοοικονομία και την συγκεκριμένη κατανομή μεταξύ των διαφόρων τομέων αυτής της βιοοικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής. Ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Θα σας ευχαριστήσω για το όσα είπανε. Συμφωνώ με την σφαιρική αυτή προσέγγιση, την οποία θα πρέπει να έχουμε και στην έκθεση αυτή και βέβαια σε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές. Και συμφωνώ κάτι το οποίο ήδη υπόθηκε, την αναγνώριση αυτή τη διαδοχική χρήση για τη βιομάζα που είχε, ήδη είχε ενταχθεί το σημείο αυτό στο κείμενο. Προφανώ η προσέγγιση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Συμφωνώ ότι όντως ε, επήγει να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε τη βιοοικονομία, γιατί πραγματικά μπορεί να αποτελέσει έναν ε, νέο τρόπο για μια νέα οικονομική ανάπτυξη και μια νέα βιομηχανική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσο με αφορά, αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνονται και τα απαραίτητα κίνητρα για την ανάπτυξη αυτής της νέας, για την ανάπτυξη αυτής της νέας οικονομίας που μπορεί να αποτελέσει μια νέα ευκαιρία για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, ως προς αυτό, θα πρέπει ε, να εγκριθεί και αυτό το παρατηρητήριο στο οποίο αναφέρθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του οποίου όντως μπορούμε πραγματικά να πιστοποιήσουμε, να επαληθεύσουμε την βιωσιμότητα της βιοοικονομίας. Η έρευνα και η ανάπτυξη είναι θεμελιώδου σημασία, αλλά είναι θεμελιώδους επίσης σημασία να υποστηρίξουμε όχι μόνο την έρευνα και την κοινωνία, αλλά να προωθήσουμε και μία ομοιομορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την βιοοικονομία, όσον αφορά τα νέα προϊόντα και τις νέες υπηρεσίες που μπορούμε να έχουμε μέσω της βιοοικονομίας ως νέο οικονομικό μοντέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά λοιπόν από αυτά που υπόθηκαν με βρίσκουν σύμφωνο. και νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε κατά αυτόν τον τρόπο μια θετική στάση και ως, τι προς τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Να ευχαριστήσω πάντως τους συναδέλφους για τη συμβολή τους για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, ευχαριστώ όλους. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική έκθεση για ένα πολύ σημαντικό θέμα. 29 Μαΐου είναι η ημερομηνία για την ψηφοφορία εδώ και προφανώς θα προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Και τώρα έχουμε το τελευταίο θέμα, το θέμα 7 κοινοτικό σύστημα καταχώρησης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών. Είναι πολύ εντυπωσιακή και η έκθεση και ο τίτλος της. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ήδη συζητήσει το θέμα αυτό εδώ στην Επιτροπή μας. Επομένως, ε, δεν θα επαναλάβω όλα όσο έχω πει για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα σταθώ στις τροπολογίες. Έκανα κάποιες τροπολογίες εγώ προσωπικά βάσει των όσων είπαμε στην πρώτη συζήτηση που κάναμε εδώ στην Επιτροπή μας. Για να σας υπενθυμίσω λίγο όμως ε, τι υπόθηκε τότε, θα σας επαναλάβω τη θέση μου. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει δηλαδή ένα ενιαίο σύστημα για την ε, καταγραφή ε, των ε, μεταφορέων ραδιενεργών υλικών, διότι αυτό αποτελεί προστιθέμενο όφελος. Θα πρέπει να πούμε ότι το καθεστώς αυτός δεν θα πρέπει να παραμείνει απλώς κενό γράμμα, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί. Και όταν το λέω αυτό, Το λέω διότι δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι αυτό θα αποτελέσει απλώς και μόνο ένα μητρό, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και μια κριτήρια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδάλλον δεν θα είναι δυνατόν να γίνεται αυτόματη αναγνώριση των πιστοποιητικών μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Κατόπιν, τι γίνεται όταν δεν γίνονται σεβαστά τα κριτήρια. Αν ένας μεταφορέας δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια, θα πρέπει αμέσως να του αποσύρεται η άδεια και να μην υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς. Και ε, κάτι επιπλέον, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό. Θα πρέπει λοιπόν ό,τι ισχύει για το σύστημα να αφορά όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να αναμερώνονται δεόντως όλα τα κράτη-μέλη για οποιαδήποτε καταχώρηση στο σύστημα. Κατόπιν, να πω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θεωρεί ως προϋπόθεση ότι τα ευρωπαϊκά όργανα είναι αλάνθαστα. Δεν υπάρχει δυνατότητα διοικητικού σφάλματος. Η Φουκουσίμα όμως μας απέδειξε ότι ακόμα και αν θεωρούμε ότι έχουμε ένα τέλειο σύστημα, πάντα υπάρχει δυνατότητα σφάλματος. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει περίπτωση να διαπιστωθούν δυσκολίες, παρατυπίες σε διοικητικό επίπεδο και επομένως θα πρέπει να προβλέψουμε και τη δυνατότητα παρέμβασης σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό όσον αφορά τις προσωπικές μου τροπολογίες. Έλαβα 60 τροπολογίες από τους πόλοιπους συναδέλφους, τους οποίους και ευχαριστώ για τις τροπολογίες τους. Στην πλειοψηφία τους οι τροπολογίες αναφέρονται στη νομική βάση η συνάδελφος Ριβαζή αναφέρεται στο θέμα του περιβάλλοντος και της υγείας. Ε, γίνεται μια αναφορά επίσης στην εσωτερική αγορά από κάποιον άλλο συνάδελφο. Πρόκειται για ε, εύστοχες παρατηρήσεις, τις οποίες θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω. Θα ήθελα να ζητήσω και την ε, άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη νομική βάση, ίσως και μια γνωμοδότηση. Υπάρχουν επίσης μια σειρά από τροπολογίε που αναφέρονται στην αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και ενιαίο, ε, εννέα κριτήρια ασφαλεία. Αυτό το αναφέρω και εγώ στις τροπολογίες μου και ε, εδώ αναφέρομαι στις ε, τροπολογίες των συναδέλφων ΠΟΚ, της κυρίας Γιανακουδάκη, η οποία αναφέρεται και ε, πως κατά πόσον επηρεάζουν αυτά τα αμοιβαία κριτήρια αναγνώρισης και τις διασυνοριακές μεταφορές. Θα ήθελα να ακούσω και για αυτά τα θέματα την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει μια τρίτη σειρά τροπολογιών. η οποία υποστηρίζει ένα ευρωπαϊκό καθεστώς μεν, αλλά θα ήθελα να επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να επιβάλλουν ε, δικά τους πρότυπα. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο σαφείς και πιο αυστηροί. Ή θα πούμε ότι δεχόμαστε ένα ευρωπαϊκό καθεστώς ή ο καθένας θα κρατήσει το εθνικό του σύστημα. Ένα μεικτό σύστημα ευρωπαϊκό και εθνικό ταυτόχρονα θα είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Θα δημιουργήσουμε ένα νέο γραφειοκρατικό τέρας το οποίο δεν θα προσφέρει τίποτα επιπλέον. Ε, Είμαι υπέρ λοιπόν ενός αμυγός ευρωπαϊκού συστήματος. Υπάρχει μία ακόμα σειρά τροπολογιών η οποία αναφέρεται σε αυτά τα ευρωπαϊκά κοινά κριτήρια Εδώ αυτά θα πρέπει να τα συζητήσω με τους σκιώδεις εισηγητές για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ ε, ανέφερα σαφώς ε, τα κριτήρια και τα έχω συμπεριλάβει στο παράρτημα, ενώ κάποιοι συνάδελφοι θα ήθελαν να συμπεριλαμβάνονται τα κριτήρια στο ε, διατακτικό. Και να ζητάτε από την, Επιτροπή, ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάζει κατάλληλες εκτελεστικές πράξεις. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, ζητώ την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, νομική βάση. Θα ήθελα να ξέρω πώς το αξιολογεί αυτή και τι γίνεται με τις επιπτώσεις των ε, κριτηρίων ασφαλείας ε, για τους πιο μικρούς μεταφορείς που διαστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και θα ήθελα να ακούσω και τις, την άποψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι τροπολογίε. Σα ευχαριστώ πολύ. Which, so, uh, headphones Βάλτε τα ακουστικά σας και θα μιλήσω την γλώσσα μου αυτή τη φορά. Σας ε, ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα και εγώ να πω ότι εξεπλάγει από τις ε, τροπολογίες κάποιες από αυτές είναι πραγματικά πάρα πολύ καλές, όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 5, που αφορούν αυτά στα οποία αναφέρομαι και εγώ με τις δικές μου τροπολογίες. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο συμφωνώ. Αν δηλαδή θέλουμε ένα ενιαίο και κοινό σύστημα, πρέπει να υιοθετήσουμε και κοινά κριτήρια. Όσο αυτά τα κριτήρια δεν είναι κοινά και ενιαία, δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί άδεια για τέτοιου είδους μεταφορά ρεδινεργών ουσιών. Αυτή είναι η άποψή μας. Θα ήθελα επίσης να εκφράσουμε με σαφήνεια τις προτεραιότητες της δικής μας πολιτικής ομάδας και αυτό το κάνουμε σε τέσσερις τροπολογίες. Συμμόρφωση με την παρούσα νομοθεσία, με την ισχύουσα νομοθεσία. Και εδώ υπάρχουν κάποιες από τις τροπολογίες μας οι οποίες ουσιαστικά συμπίπτουν με την εισηγήτρια των Πρασίνων και τις τροπολογίες της. Θα ήθελα επίση να πω ότι αν όντως υπάρχει πληροφόρηση όσον αφορά την συμβατότητα, τη συμμόρφωση αυτή θα πρέπει να κοινοποιείται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Και από τη στιγμή που υπάρχει συμμόρφωση τότε θα δίνεται άδεια για μεταφορά. Βεβαίω, κάποιες από τι τροπολογίε ε, των πασίνων μπορούμε να τις υποστηρίξουμε άμεσα, κάποιε, θα πρέπει να τις συζητήσουμε περαιτέρω και θα ήθελα να ακούσω βεβαίω και την Επιτροπή γιατί εδώ δεν ξέρουμε ακριβώ ποια θα είναι η νομική βάση. Όσον αφορά την τροπολογία που αφορά την εθνική νομοθεσία, η οποία θα πρέπει να προέχει της ε, ευρωπαϊκής, αν υιοθετήσουμε μια τέτοια προσέγγιση, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε κοινοτική και ενιαία νομοθεσία. Πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Βλέπω ότι μπορεί να γίνουν πολλοί συμβιβασμοί και βεβαίως θα συνεχίσω να επεξεργάζομαι το κείμενο με την εισηγήτρια. Η κυρία Γιάννα Κουδάκη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη. Εν γέννη συμφωνούμε με τον εισηγητή και την έκθεσή του. Νομίζουμε ότι είναι καλή και είναι σαφώ θετικό το ότι απλουστεύουν διαδικασίε για τι επιχειρήσει. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό για τις επιχειρήσεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μεταφορέα. Υπάρχουν καλές σχετικές διακάσεις στον κανονισμό. Το να έχουμε πλέον ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα καταχώρησης ε, για το τομέα των μεταφορών. Αυτό είναι θετικό γιατί μπορεί να οδηγήσει τελικά σε ελάφρυνση του διοικητικού άχθους, καλύτερη εναρμόνιση. Και μου αρέσει ιδιαίτερα το το κείμενο είναι ιδιαίτερα στεναρό στο σημείο αυτό. Δηλαδή ότι όταν κάποιο δεν συμμορφώνεται, αυτό κοινοποιείται προ τα έξω. Αυτό είναι σαφέ δείγμα διαφάνεια. Έπειτα, νομική βάση. Πάρα πολλοί αναφέρθηκαν σε αυτό. Δεν υπάρχει λόγο να επεκταθώ περισσότερο. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ρωτάω και εγώ, να μα πει ποια είναι η άποψή τη. Η κυρία Γκροστέτ έχει το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκροστέτ πρώτη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη. Ήδη συζητήσαμε την έκθεση αυτή και στο παρελθόν, η κυρία Τζόρνταν. Προσπάθησε να συντάξει μια ισορροπημένη έκθεση. Νομίζω ότι η προσπάθεια της αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Απλώς έχω κάποιες αμφιβολίες γιατί νομίζω ότι μέσω της έκθεσης αυτής προσπαθούμε ουσιαστικά να αναφερθούμε σε πρώτερες διατάξεις ε, της συνθήκης Ευρατόμ και κάπως αυτό με ενοχλεί. Το είχα πει και στην κυρία Τζόρνταν ότι δεν συμφωνούσα απολύτω με όλε τι τροπολογίε τη. Ε, Ορισμένε τι έβρισκα κάπω προβληματικέ. 3, 3, 10 και 13. Δεν συμφωνώ με τι τρει αυτέ τροπολογίε γιατί υπάρχουν ήδη νομοθετικέ πράξει που αναφέρονται στα σημεία αυτά και που αναφέρονται άλλωστε και στην έκθεσή τη. Επομένως, η αρχή της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών θα πρέπει να διατηρηθεί. Τροπολογία 6. Νομίζω ότι είναι κάπως υπερβολική δυνατότητα του ε, κράτους μέλους ε, να λαμβάνει δράση σε σχέση με το κράτος μέλος εκείνο το οποίο αποστέλει τα εμπορεύματα και τροπολογία 7 στη συνέχεια τη θεωρώ κάπως περιττή. Και νομίζω ότι εν τέλει δίνουμε πολλές αρμοδιότητες εκτελεστικές στην Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και αυτό κάπως με ενοχλεί. Δεν θα, να αναφερθώ τώρα στις τροπολογίες της κυρίας Ριβαζή, η οποία θέλει να αλλάξει μέσω τροπολογιών της την ε, νομική βάση του κειμένου. Μας έχει συνηθίσει σε τέτοια, στάση. Εγώ αυτό που θέλω να της πω και να πω σε όλους είναι ότι έχουμε τη συνθήκη Ευρατόμ, ας επαληθεύσουμε ότι όντω εφαρμόζονται καλά οι οδηγίες που πορεύουν από τη συνθήκη αυτή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βάλουμε κατά τη συνθήκη σε βρατών κάθε φορά που μας δίνει τη ευκαιρία. Αυτό με ενοχλεί όλους ιδιαίτερος. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Μου είπατε αρκετές φορές να σας πω κάτι για τη νομική βάση. Να σας υπενθυμίσω ότι το 2002 υπήρξε μια απόφαση στο δικαστηρίου, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο φυσικά, η οποία αναφέρθηκε στην εξουσία που δίνεται από το κεφάλαιο 3, ε, άρθρο 30, 32, ε, αυτό το οποίο προτείνουμε και εμείς ως νομική βάση και υπενθυμίζω ότι είπε το Ευρωπαϊκό ε, δικαστήριο. Το δικαστήριο αναγνωρίζει ότι τα άρθρα 30 και 32 προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευρεία νομοθετική αρμοδιότητα για θέματα προστασίας της υγείας και για το σύστημα ε, πιστοποίησης, αυτό που προτείνουμε εδώ, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη. Η νομοθετική αυτή πράξη αποτελεί ένα συμπληρωματικό μέτρο για τη ε, πρότυπα ασφαλείας. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει αυτό το οποίο είχαμε και εμείς στο σχέδιο κανονισμού. Η άποψή μας λοιπόν είναι ότι ε, αυτή είναι η σωστή νομική βάση, τα άρθρα 30-32 της ε, συνθήκης. Τώρα, ε, την άποψή μας για τα κριτήρια, να σας πω ότι εμείς θα υποστηρίξουμε και υπήρχε, υπάρχει μια ανάλογη πρωτοβουλία στο ε, Συμβούλιο για να υπάρχει ένα παράρτημα με τα κριτήρια, την αναφορά λοιπόν σε κριτήρια αυτά και θα δούμε κατά πόσον είναι δυνατόν να συμπεριλάβουμε και αυτά τα κριτήρια. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου η οποία θα αναφέρει στην Προεδρία πώς ε, μπορούν να τροποποιήσουν τον κανονισμό ώστε να είναι ακόμα πιο στεναρός και αυτό φυσικά πηγαίνει ακριβώς και ε, προς την κατεύθυνση αυτών που προτείνει η συντάκτρια της νομοδότησης. Να έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια ε, εμείς ε, προτείνουμε να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, αλλά να μην είναι τόσο διεξοδικές οι αναφορές όπως ε, προτείνει η συντάκτηρα της νομοδότησης. Αλλά επειδή ακριβώς προτείνετε κι εσείς ακριβώς το ίδιο με το Συμβούλιο, θα το επεκτείνουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ, συγγήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τα σχόλιά τους και εγώ θα ήθελα να μας δώσετε αυτό το έγγραφο που αναφέρεται στη νομική βάση. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα αυτό, σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούμε την συνθήκη Euratom. Το μόνο που θα ήθελα να κάνω είναι να διευκρινίσουμε τη νομική βάση και ευχαριστώ όλους για τα σχόλια. Θα συνεργαστούμε με τους και όδησης για να βρούμε κοινέ προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ενδεικτικά σας λέω ότι έχουμε προβλέψει ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Τελειώσαμε για σήμερα. Θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί στις 10 και με την ψηφοφορία. Έχουμε τα ελαφρά εμπορικά οχήματα αύριο. Σας παρακαλώ πολύ να είσαστε ακριβείς για την ψηφοφορία.